Το ραντεβού μας ήταν στις 3 ακριβώς. Αφήσαμε ένα ακαδημαϊκό δεκάλεπτο από αυρότητα, αλλά νομίζω ότι είναι ώρα να ξεκινήσουμε την απογευματινή μας συνεδρίαση με το σημείο 9 της ημερήσιας διάταξης που προβλέπει συζήτηση για την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Εσωτερικής Ασφάλειας. Θα ακούσουμε την παρέμβαση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ΚΟΖΗ, τη μόνιμη επιτροπή για θέματα συνεργασία και εσωτερικές ασφάλειες και την εισηγήτριά μας την κυρία Μπορσελίνο. Θα θυμάστε ότι στη τελευταία διάσκεψη που έγινε την 5η ε, Οκτωβρίου ε, για το θέμα αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξήγηλε την πρώτη ε, αυτή η έκθεση και μάλιστα ακούσαμε τις πρώτες πληροφορίες από την ΚΟΖΗ, την ε, μόνιμη επιτροπή. Τώρα έχουμε λάβει στο μεταξύ την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θέλουμε τις συμπληρωματικές πληροφορίες του Συμβουλίου από την Επιτροπή Εσωτερικής Ασφάλειας. Αυτή θα αποτελέσει και τη βάση την έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας που ε, θα εκπονήσει η κυρία Μπορσελίνο και που θα συμπληρώσει το έργο της κυρίας Αλφάνο για το οργανωμένο έγκλημα και της κυρίας Χίνμπελτ για την εξολόγηση των προσπαθειών πάταξης δρομοκρατίας. Πρώτα θα δώσω το λόγο στον κύριο Μύροσλαφ Κομάνεκ, τον οποίο και καλωσορίζω και που είναι αντιπρόεδρος της ΚΟΖΗ, της Επιτροπής Εσωτερικής Ασφάλειας. αν δεν κάνω λάθος, είναι εδώ και ο κύριος Νούνες Δελμέιντα, εκπροσωπώντας την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα μας ενημερώσουν για τις εξελίξεις. Πρώτα λοιπόν έχει το λόγο ο κύριος Μύροσουαφ Κουμάνεκ. Σας ακούμε. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμοι Ευρωβουλευτέ, κυρίες και κύριοι, εκ μέρους του Πρόεδρου της ΚΟΖΗ, του κυρίου Ριπάλτσκη, που δυστυχώς ε, ε, χρειάστηκε να μεταβεί σε κατεπίγουσα αποστολή στην Πολωνία, θα σας ενημερώσω εγώ αναπληρώνοντάς το για τις εξελίξεις της Ευρωπαϊ... των ευρωπαϊκών προσπαθειών σε τη φορά την πάταξη οργανωμένου και σοβαρού εγκλήματος. Η η μόνιμη επιτροπή για συνεργασία και εσωτερική ασφάλεια, που είναι γνωστή και ως επιτροπή ΚΟΖΗ, ε, θεσπίστηκε προκειμένου να διευκολύνει, να προωθήσει και να ενισχύσει την ε, επιχειρησιακή συνεργασία των αρμόδιων εθνικών αρχών των ευρωπαϊκών χωρών σε θέματα εσωτερικής ασφάλειας. Έργο της μόνιμης αυτής επιτροπής είναι να εξασφαλίσει μια αποτελεσματική συνεργασία και συντονισμό σε θέματα συνεργασίας αστυνομικής και τελωνιακής και σε αρμοδιότητες και σε επιχειρήσεις ελέγχου εξωτερικών συνόρων. Η μόνιμη αυτή επιτροπή θα αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων και της συνεργασίας, θα εντοπίσει ενδεχόμενες αδυναμίες και στη συνέχεια θα προτείνει δράσεις προκειμένου να καλυφθούν και να διορθωθούν οι αδυναμίες. Η μόνιμη αυτή επιτροπή, η ΚΟΖΗ, δεν συμμετέχει στην διεξαγωγή επιχειρήσεων ή στην εκπόνηση νομοθετικών πράξεων. Η μόνιμη αυτή επιτροπή συμβάλλει και στην εξασφάλιση συνοχής των δράσεων της Eurojust, της Europol, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Εξωτερικών Συνόρων, Frontex δηλαδή, και άλλων ε, σχετικών οργάνων. Όλα αυτά τα όργανα συμμετέχουν ως παρατηρητές στις συνεδριάσεις της μόνιμης αυτής Επιτροπής Εσωτερικής Ασφάλειας, της COSI. Ο κύκλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για οργανωμένο και σοβαρό έγκλημα προβλέπονται στα συμπεράσματα του, του Συμβουλίου Εξωτερικών, Εξωτερικών Υποθέσεων του 2010 προκειμένου να αντιμετωπιστούν με μεθοδολογικό και πιο συνεπή τρόπο οι διάφορες απειλέ, χάρη στην βέλτιστη συνεργασία μεταξύ των αρμοδίων υπηρεσιών των κρατών μελών, των κοινοτικών θεσμικών οργάνων και των ε, κοινοτικών οργανισμών καθώς και ενδιαφερόμενων τρίτων χωρών και άλλων διεθνών οργανώσεων. Ε, τέσσερις είναι οι φάσεις του Ευρωπαϊκού Κύκλου Πολιτικών. Η πρώτη φάση είναι η ε, ε, ανάπτυξη, σχεδιασμός των πολιτικών με βάση αξιολόγηση των απειλών από οργανωμένο και σοβαρό έγκλημα. Χάρη στην μελέτη αυτή θα γίνει μια επισκόπηση των απειλών κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η δεύτερη φάση του κύκλου είναι ε, ο σχεδιασμός πολιτικής, η διαμόρφωση πολιτικής και η λήψη αποφάσεων ε, ε, και ο περιορισμός από το Συμβούλιο συγκεκριμένων προτεραιοτήτων σε περιφερειακό και πανευρωπαϊκό επίπεδο. Για κάθε προτεραιότητα προβλέπεται ένα πολιετές στρατηγικό σχέδιο προκειμένου να εξασφαλιστεί ένας ε, ε, διακλαδικός και ολοκληρωμένος τρόπος κάλυψης των μέτρων αυτών προκειμένου να αντιμετωπιστούν δεόντως ε, οι απειλές με βάση την ιεράρχηση που έχει γίνει. Η τρίτη φάση αφορά την εφαρμογή και παρακολούθηση του ετήσιου επιχειρησιακού σχεδίου δράσης που ευθυγραμμίζεται φυσικά με τους στρατηγικούς στόχους όπως προβλέπονται στο πολιετές σχέδιο στρατηγικής και λαμβάνει υπόψη το σχέδιο της Κοσπόλ που θα είναι το πολυμερές πρέσιο για την αντιμετώπιση των απειλών όπως έχουν ιεραρχηθεί και ο τέταρτος κύκλος, η τέταρτη φάση του κύκλου πολιτικής είναι μια ενδελεχής αξιολόγηση κατά το τέλος του κύκλου που θα αποτελέσει σημαντικό input ε, για την προετοιμασία του επόμενου κύκλου. Το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο αρχικός διετής κύκλος πολιτικής θα εφαρμοστεί για την περίοδο 2011 έως 2013 με βάση την αξιολόγηση απειλών από οργανωμένο έγκλημα του 2011. Με βάση την αξιολόγηση του αρχικού κύκλου της πολιτικής προβλέπεται ένας τετραετής κύκλος εφαρμογής που θα καλύψει την περίοδο 2014 έως 2013-2017 με βάση την ε, αξιολόγηση ε, για τις απειλές από σοβαρό και οργανωμένο έγκλημα το 2013. Η ΚΟΖΗ έλαβε την εντολή από το Συμβούλιο να υποβάλει ε, επί τη βάση του Συμβουλευτικού Οργάνου Πολιτικής ε, που συνέταξαν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Προεδρία και στηριζόταν στο ΟΚΤΑ το 2009 και την ε, Ευρωπαϊκή ΣΟΚΤΑ του 2013 και έπειτα κάποια συμπεράσματα προς το Συμβούλιο με προτεραιότητες και προτάσεις για το πολιτές ε, στρατηγικό σχέδιο καθώς και για τα επιχειρησιακά ετήσια σχέδια προκειμένου να γίνει σωστή παρακολούθηση και επίβλεψη αυτής της εφαρμογής. Αναγνωρίστηκε φυσικά η σημασία των βασικών προκλήσεων που ε, περιλαμβάνει αυτή η στρατηγική εσωτερική ε, ασφάλειας, αλλά ο κύκλος πολιτικής εστιάστηκε κυρίως σε σοβαρό και οργανωμένο έγκλημα. Τον Ιούνιο του 2011 το Συμβούλιο ε, έχει ως προτεραιότητα καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος για την περίοδο 2011 με 2013 ε, και μάλιστα οι προτεραιότητες αυτές ε, είναι οκτώ με πρώτη την αποδυνάμωση των οργάνων, των ομάδων οργανωμένων εγκλήματος που έχουν έδρα στη Δυτική Αφρική ε, και που ασχολούνται με λαθρεμπόριο ναρκωτικών, ηρωίνης και κοκαίνης από και προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η δεύτερη προτεραιότητα, μετριασμός ε, του ρόλου των ε, Δυτικών Βαλκανίων ως βασική ζώνη διέλευσης και αποθήκευσης για παράνομα προϊόντα με προορισμό την Ευρωπαϊκή Ένωση και επιμελητιακό κέντρο για οργανωμένα κυκλώματα εγκλήματος συμπεριλαμβανομένων αλβανόφωνων συμμοριών οργανωμένου εγκλήματος. Τρίτη προτεραιότητα. Αποδυνάμωση του, της ικανότητας οργανωμένων ομάδων εγκλήματος να προωθούν λαθρομετανάστες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίως μέσω των νοτίων, της νότιας, νοτιοανατολικής και ανατολικής Ευρώπης και κυρίως στα ελληνοτουρκικά σύνορα και σε περιοχές κρίσης της Μεσογείου κοντά στην Βόρεια Αφρική. Επόμενη προτεραιότητα. Η μείωση της παραγωγής και διανομής συνθετικών ναρκωτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συμπεριλαμβανομένων και νέων ε, ψυχοδραστικών ουσιών και ψυχότροπων φαρμάκων. Άλλη προτεραιότητα είναι διατάρα, αναχέτηση του εμπορίου παράνομων προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως κοκαίνη, ηρωίνη, κάναβης, παραποιημένα προϊόντα ή απομίμησης και ε, σιγαρέτα. Άλλη προτεραιότητα του Συμβουλίου είναι η καταπολέμηση πάσης ε, μορφής ε, εμπορίου ανθρώπων προκειμένου να εξαρθρωθούν ε, τέτοιες συμμορίες οργανωμένα εγκλήματος, ιδιαίτερα στους ε, νότιους και νοτιοανατολικούς, καθώς και ανατολικούς κόμβους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άλλος στόχος είναι η μείωση της, του, της γενικής ικανότητας κινητών ομάδων οργανωμένου εγκλήματος για διάπραξη τέτοιων εγκληματικών δράσεων και τελευταία προτεραιότητα είναι η αναβάθμιση του αγώνα κατά το εγκλήματος στον κυβερνοχώρο και η αποφυγή της κατάχρησης του, του κυβερνοχώρου από εγκληματικές ομάδες. Η ΚΟΖΗ ανέλαβε την προσπάθεια συντονισμού, παρακολούθηση και αξιολόγηση τη εφαρμογή των στρατηγικών στόχων και των ετήσιων επιχειρησιακών σχεδίων δράση για κάθε προτεραιότητα. Επίσης, ε, η ΚΟΖΗ εξασφαλίζει τη συνεπή εφαρμογή των διαφόρων επιχειρησιακών δράσεων που είναι απαραίτητες για την ενίσχυση της εσωτερικής ασφάλειας ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων εθνικών αρχών και των ε, κοινοτικών ενωσιακών οργανισμών. Η ΚΟΖΗ ανέλαβε την εντολή από το Συμβούλιο προκειμένου να εξασφαλίσει οι δράσεις που εφαρμόζονται κατά οργανωμένου και σοβαρού εγκλήματος να είναι συνεπείς με τους στρατηγικούς στόχους που θα υιοθετήσει η ΚΟΖΗ και, τις ε, και τα επιχειρησιακά σχέδια δράσης που θα εγκρίνει. Μεταξύ Ιουλίου και Οκτωβρίου 2011 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την υποστήριξη της Φοροεδρίας και της Europol οργάνωσε σεμινάρια για κάθε μία προτεραιότητα χωριστά με συμμετοχή χωρών μελών και εμπειρογνωμόνων από τους κοινοτικούς οργανισμούς προκειμένου να εκπονηθούν οι στρατηγικοί στόχοι για κάθε προτεραιότητα. Μάλιστα, με βάση τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σε ό,τι αφορά την ε, δημιουργία και εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κύκλου Πολιτικής. Στην αρχική διετή φάση του κύκλου θα θεσπιστούν κάποιοι στρατηγικοί στόχοι πριν την υποβολή του πολιτούς ε, στρατηγικού σχεδίου. Τέτοια ε, στρατηγικά σχέδια προβλέπονται στον τετραετή κύκλο πολιτικής. Οι στρατηγικοί στόχοι υποβλήθηκαν κατόπιν στην Επιτροπή Κόζη που τους ενέκρινε στις 8 Σεπτεμβρίου. Τον Οκτώβριο του 2011 η Europol οργάνωσε σεμινάρια με στόχο την, την εκπόνηση των ετήσιων επιχειρησιακών σχεδίων δράσης για κάθε προτεραιότητα χωριστά με βάση τους στρατηγικούς στόχους που, είχαν, που είχε νωρίτερα ε, καταρτήσει η Επιτροπή Κόζη. Το έργο για αυτά τα ετήσια επιχειρησιακά σχέδια δράσης έχει ολοκληρωθεί μόλις πρόσφατα και τα σχέδια αυτά θα υποβληθούν στην Επιτροπή Κόζη προς έγκριση τον Δεκέμβριο. Μετά την έγκριση αυτών των, την επικύρωση αυτών των ετήσιων σχεδίων ε, δράσης θα περάσουν στις αρχές του 2012 σε ε, φάση εφαρμογής. Η ΚΟΖΗ θα παρακολουθήσει το, την πρόοδο κάθε, ανά εξάμεινο κάθε ε, ετήσιου επιχειρησιακού σχεδίου δράσης. Και μάλιστα υπάρχει και μία πολυμερής πλατφόρμα για την συζήτηση και τον εντοπισμό των απειλών κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχει τα αρχικά impact. Ε, θα συστηθεί αυτή η πολυμερής ε, πλατφόρμα στα πλαίσια του ισχύοντος ε, σχεδίου COSPA και επίσης θα παρακολουθεί την εφαρμογή των ετήσιων επιχειρησιακών σχεδίων δράσης και το έργο για τη διαμόρφωση, για την οριστικοποίηση της πλατφόρμας αυτής συνεχίζεται. Τα επιχειρησιακά μέτρα που θα εφαρμοστούν στα πλαίσια της ευρωπαϊκής πολιτικής θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη στους διάφορους τομείς δραστηριοτήτων και την εξωτερική διάσταση της ε, εσωτερικής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και το θέμα του εντοπισμού και της ε, κατάσχεσης δίμευσης ε, περιουσιακών στοιχείων εγκληματικών οργανώσεων. Και στα πλαίσια του κοινού εγγράφου για την ενίσχυση των δεσμών στα πλαίσια της κοινή ε, εξωτερικής πολιτικής ε, ε, και πολιτικής άμυνας καθώς και του Ευρωπαϊκού Χώρου Ασφάλειας και Δικαιοσύνης, η ΚΟΖΗ έχει ξεκινήσει πολιτικό διάλογο με την Πολιτική Επιτροπή και Επιτροπή Ασφάλειας προκειμένου να εντοπιστούν τομείς συνεργασίας και να γίνει μια σύσφυξη της συνεργασίας των δύο αυτών επιπέδων. Συνεχίζεται μάλιστα ο διάλογο της ΚΟΖΗ με τις, με τις δύο αυτές ε, επιτροπές. Φυσικά, στόχος της ΚΟΖΗ είναι να αποτραπεί και να ε, καταπολεμηθεί το οργανωμένο έγκλημα με βάση τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για τις κινητές ομάδες οργανωμένου εγκλήματος του Δεκεμβρίου του 2010 και έτσι διευρύνθηκε το άτυπο δίκτυο αξιωματοχών επαφής προκειμένου να καλύπτει το δίκτυο αυτό και άλλα φαινόμενα σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος, όπως καθορίζονται από τις ευρωπαϊκές προτεραιότητες και περιλαμβάνονται στον ευρωπαϊκό κύκλο πολιτικής. Ο Ευρωπαϊκό Κύκλο Πολιτική για το Οργανωμένο και Σοβαρό ε, Έγκλημα είναι ένα μοναδικό εργαλείο και μάλιστα είναι και ένα καινοτόμο εργαλείο άνευ προηγουμένου γιατί μεταμορφώνει τις πολιτικές προτεραιότητες σε συγκεκριμένες και απτές δράσεις, θεσπίζοντας μια σαφή μεθοδολογία για την διαμόρφωση, εφαρμογή και αξιολόγηση προτεραιοτήτων στην καταπολέμηση σοβαρού και οργανωμένου διεθνούς εγκλήματος και μάλιστα με έναν συνεκτικό, διακλαδικό και ολοκληρωμένο τρόπο που συμβάλλει στην αύξηση της αξιοπιστίας, της λογοδοσίας, της αποτελεσματικότητας και της συνοχής των δράσεων. Αξιότιμη Ευρωβουλευτέ, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την προσοχή που δώσατε και να σας διαβεβαιώσω ότι είμαι στη διάθεσή σας για να λύσω τις απορίες σας. Όχι, εμείς σας ευχαριστούμε κύριε Κουμπάνεκ. Τώρα η εκπρόσωπος της Κομισιόν κύριος Λούνες Δαλμέιδα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Αγαπητοί Ευρωβουλευτέ, είναι μεγάλη μου τιμή που προσεκλήθην στην Επιτροπή σας για να σας εξηγήσω την πρώτη ετήσια έκθεση της Κομισιόν για την εφαρμογή της στρατηγικής που αποφασίστηκε την περασμένη Παρασκευή. Πέρυσι, όπως γνωρίζετε, η Κομισιόν ενέκρινε μια ανακοίνωση για το θέμα της εσωτερικής ε, στρατηγικής ασφαλείας της Ένωσης που αντιπροσωπεύει το κοινό πρόγραμμα των χωρών και του Κοινοβουλίου για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που μας περιμένουν από το 10 μέχρι το 14. Γι' αυτόν τον σκοπό ταύτισε η ανακοίνωση πέντε προτεραιότητες όπου μπορεί πράγματι να προσφέρει κάτι η Κομισιόν και να προτείνει συγκεκριμένη δράση. Κατά πολέμηση και πρόληψη του οργανωμένου εγκλήματος ήταν το πρώτο, δεύτερον τρομοκρατία τρίτον κυβερνοέγκλημα, τέταρτον ενδυνάμωση της διαχείρισης των εσωτερικών συνόρων και πέμπτον, πέμπτον λέγω, αντιμετώπιση θεομηνιών για να οικοδομηθεί μια ανοιχτή αλλά και ασφαλής Ευρώπη όπως προέβλεπε το πρόγραμμα της Στοκχόλμης συμβουλευτήκαμε στοιχεία που έδειχναν ότι και οι πέντε αυτές προκλήσεις είναι σημαντικές για την εσωτερική ασφάλεια της Ένωσης. Πολλοί Ευρωπαίοι και Ευρωπαίες πιστεύουν επίσης ότι οι απειλές που προκύπτουν από, αυτά τα πέντε, από αυτές τις πέντε προκλήσεις θα αυξηθούν και γι' αυτό θελήσαμε σε συνεργασία με όλες τις υπηρεσίες της Ένωσης να δούμε πώς μπορεί να εφαρμοστεί η καταπολέμηση των πέντε προκλήσεων. Ένα χρόνο μετά είναι πια καιρός να δούμε τι πετύχαμε ως προς την εσωτερική ασφάλεια και για τους πέντε στόχους. Τι πετύχαμε το 11? Το 11 υπήρξε υποσχόμενο έτος για την εφαρμογή της στρατηγικής αυτής, αλλά οι απειλές του Νοεμβρίου 10 δεν ε, σταμάτησαν. Δηλαδή, για κάθε μία από τις πέντε προτεραιότητες που είχαμε ταυτίσει πέρυσι μπορούμε να αναφέρουμε την εξής πρόοδο. Πρώτον, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Σημαντική πρόοδος έχει επιτευχθεί το 2011. Ιδιαίτερα ως προς την πρότασή μας για ενωσιακή νομοθεσία για συλλογή στοιχείων των επιβατών που μπαίνουν και βγαίνουν από την Ένωση. Χρειάζεται όμως περαιτέρω πρόοδος για τη συνεργασία των διοκτικών αρχών και για να αναπτυχθεί καλύτερη διοικητική συνεργασία στην καταπολέμηση του οργανωμένου κλίματος. Για την τρομοκρατία και τη ριζοσπαστικοποίηση των λαών χρειάστηκε να δημιουργήσουμε ολόκληρο δίκτυο και η έγκριση ειδική δήλωση ή ανακοίνωση της Κομισιόν για το θέμα αυτό αποτελεί επίσης ένα σημαντικό βήμα. Όσο για τα διοικητικά μέτρα για το πάγωμα λογαριασμών τρομοκρατών και τρομοκρατριών, η έκθεσή μας τονίζει ότι χρειάζονται και εδώ περαιτέρω προσπάθειες. Η δράση καταπολέμησης του κυβερνοεγκλήματος έχει προχωρήσει και σημειωθεί πρόοδος για τη δημιουργία ενός πανενοσιακού κυβερνοεγκληματικού κέντρου. Με συγχωρείτε, έχω κρυώσει. Η Κομισιόν καλεί τα κράτη-μέλη να αναλάβουν επίγουσα δράση για να εφαρμόσουν τη σύμβαση της Βιδαπέστης. Ως προς τη διαχείριση και έλεγχο των συνόρων, συζητιέται ακόμη η εφαρμογή αυτού του ευρωπαϊκού συστήματος για τα σύνορα, για τους ελέγχους στα σύνορα. Πρέπει όμως και εδώ να υπάρξει πρόοδος. Για τη διαχείριση κρίσεων και καταστροφών και θεομηνιών επίσης κάτι έχουμε κάνει. Το 11 παραδείγματος χάρη για την αξιολόγηση κινδύνων. Αλλά και εδώ τονίζουμε ότι χρειάζονται περαιτέρω προσπάθειες. Επίσης τονίζουμε ότι έγιναν μερικά βήματα το χάσμα μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών πτυχών της ασφαλείας της Ένωσης. Υπήρξαν, ανελήφθησαν πολλές πρωτοβουλίες για καλύτερο συντονισμό όπως πρακτική συνεργασία αντιτρομοκρατικών οργανώσεων και έλεγχο της παράνομης μετανάστευσης από τα Δυτικά Βαλκάνια, τη Σαχάρα κλπ. Υπήρξε ένα κοινό έγγραφο, είπα και... Ε, για την ασφάλεια και τη συνεργασία μεταξύ άλλων τονίσαμε ότι χρειάζεται καλύτερη συνεργασία μεταξύ Ευρωπόλ και μεμονωμένων αστυνομικών δυνάμεων. Τι άλλο πρέπει να γίνει. Και στους πέντε τομείς ταυτίσαμε τις ανάγκες και τις απειλές όπως που προκύπτουν μάλλον από την πολύ γρήγορη πρόοδο της λειτουργίας και επέκτασης του διαδικτύου που θέτει καινούρια προβλήματα ασφαλείας. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει η Ένωση να είναι ανοιχτή σε περαιτέρω πρόοδους και γι' αυτό θελήσαμε να ταυτίσουμε τι πρέπει να γίνει το 12 τι δράσεις πρέπει να αναλυφθούν και από εμά και από τα κράτη-μέλη μεμονωμένα. Και εδώ χρειάζεται περαιτέρω πρόοδος, ιδίως ως προς την καταπολέμηση του οργανωμένου και σοβαρού εγκλήματος, αλλά και του κυβερνού εγκλήματος επί του οποίου θα αναφέρω μερικές λεπτομέρειες. Για την καταπολέμηση του βαρού και οργανωμένου εγκλήματος αυτό που πρέπει να γνωρίζουμε είναι ότι δημιουργείται αυτή τη στιγμή ένας νέος εγκληματικός χώρος και δημιουργούνται εγκληματικές ομάδες πολύ πιο ευέλικτες από ό,τι πριν οι οποίες βοηθούνται από την διαδεδομένη χρήση του ίντερνετ. Δημιουργούνται όλο και περισσότερες τρομοκρατικές και εγκληματικές ομάδες οι οποίες ε, ε, συνδέονται διότι το οργανωμένο έγκλημα χρηματοδοτεί πολλές φορές την τρομοκρατία. Ένα από τα κυριότερα στοιχεία για να αντιμετωπιστεί αυτή η πρόκληση κατά πολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος είναι η διαμεθοριακή συνεργασία και η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εθνικών αρχών. Παρ' όλα αυτά, η ενωσιακή νομοθεσία, ιδιαίτερα η Σουηδική πρωτοβουλία, δεν έχει ακόμη εφαρμοστεί από τα κράτη-μέλη. Επίσης λυπούμαστε διότι τα διάφορες υπηρεσίες μέσα και εργαλεία που έχουν προβλεφθεί δεν έχουν ακόμη πλήρως επικυρωθεί από όλες τις χώρες μέλη. Πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι θα υπάρξει μία πιο αποτελεσματική συνεργασία στον τομέα των διώξεων. Τέλος θα ήθελα να τονίσω τι πρέπει να γίνει για να παγώνουν και να κατάσχονται πιο αποτελεσματικά και πιο γρήγορα οι λογαριασμοί των εγκληματιών και τα περιουσιακά των στοιχεία. Οι εγκληματίες πολλές φορές ζητούν, θέλουν να επενδύουν τα παράνομα κέρδη τους σε νόμιμες δραστηριότητες, αυτό που λέμε ξεπλήμα βρωμίκου χρήματος δηλαδή. Τι θέλουμε λοιπόν, τι πρέπει να κάνουμε το 12 για να ανταποκριθούμε σε αυτές τις προκλήσεις. Θα προτείνουμε μία δέσμη για τις κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων κλιματιών, πρόταση για τη μεταρρύθμιση της λειτουργίας της Ευρωπόλ, Ευρωτζάστ και ΣΥΠΟΛ, καθώς και την πρόσληψη περισσότερων επαγγελματιών. Θα υποβάλουμε προτάσεις για οδηγίες καταπολέμησης του ξεπλήματος βρωμίκου χρήματος και με βάση τις αποφάσεις Προύβ και της Σουηδικής Πρωτοβουλίας θα ζητήσουμε ένα νέο πρότυπο ανταλλαγής πληροφοριών. Τώρα για το κυβερνοέγκουλημα. Και αυτό αυξάνεται και μεγάλος στόχος του είναι η Ένωση λόγω του γεγονότος ότι έχει διαδεδομένα δίκτυα χρηστών διαδικτύου. Επειδή έχει προχωρήσει πολύ η τεχνολογία αυξάνεται και το κυβερνοέγκλημα. Η χρήση όλο και περισσότερων cloud computing δηλαδή που μπορεί σε περίπτωση επίθεσης να ζημιώσει πολύ περισσότερο τους χρήστες. Επίσης σημειώθηκε πολύ μεγάλη αύξηση των εγκλημάτων κατά των δικαιωμάτων, πνευματικών δικαιωμάτων, παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων. Πολλοί θεωρούν ότι το κυβερνοέγκλημα σταματάει στα εθνικά σύνορα, αλλά δεν ισχύει αυτό. Πρέπει να μπορούμε να είμαστε σε θέση να έχουμε μια κοινή ανταπόκριση, απάντηση σε, τέτοια, σε τέτοιες επιθέσεις. Το 12 λοιπόν θα θέλαμε να οργανωθεί μια τέτοια στρατηγική δικτύωση μέσω της οργάνωσης ενός κέντρου καταπολέμησης του κυβερνοεγκλήματος πανενωσιακού. Και το ίδιο θα συζητήσει και η ομάδα ήπα ΕΠΑ-ΕΕ. Οι Πολωνοί συνάδελφοί μας τόνισαν έκαναν μάλλον ως Προεδρία προτάσεις τις οποίες δεχόμαστε πλήρως και η εφαρμογή των στόχων της εσωτερικ... στρατηγικής εσωτερικής ασφαλείας θα συνεχίσει αλλά δεν θα αρκέσει. Πρέπει όλα αυτά να μεταφραστούν σε δράση και γι' αυτό όπως σας είπα η Κομισιόν δέχεται τη μεθοδολογία αυτού του κύκλου που πρότεινε η Πολωνική Προεδρία για την καλύτερη εκτίμηση και οργάνωση των απειλών που σημειώνονται μεταξύ άλλων και στο κυβερνοέγκλημα και υποστηρίζουμε πλήρως τα συμπεράσματα του Συμβουλίου του Ιουνίου του 2011 που, τις πέντε αυτές, που εγκρίνουν τις πέντε αυτές προτεραιότητες μέχρι και το 2013. Τελεία. Με την στρατηγική αυτή ασφαλείας και τον κύκλο πολιτικής της Ένωσης δεσμευτήκαμε να εφαρμόσουμε μια συνεπή πολιτική με σαφείς προτεραιότητες. Και ο αντιπρόεδρος του Κόζη σας ανέφερε ήδη τις νεότερες πληροφορίες ως προς το τι συζητιέται εκεί γιατί νομίζουμε ότι και η Κόζη μπορεί να δημιουργήσει σοβαρή ορμή για πρόοδο. Κύριες και κύριοι βουλευτέ, τώρα πρέπει το ρόλο του να τον παίξει και το Κοινοβούλιο γιατί είναι πολύ σημαντικός και εμείς προσπαθήσαμε να σας δώσουμε ό,τι πληροφορίες χρειάζοσασταν. Μεταξύ άλλων αυτή η ετήσια έκθεση ελπίζουμε να αποτελέσει τη βάση για τις αναλύσεις και τις αποφάσεις σας διότι θα θέλαμε και το Κοινοβούλιο να εγκρίνει αυτή τη στρατηγική στην έκθεση Μπορσαλίνο. που ελπίζουμε να συμπεριλάβει όλα μας τα συμπαράσματα στην έκθεση ιδίας πρωτοβουλία της. Όπως είπα το 11 ήταν μια πολλά υποσχόμενη αρχή αλλά μένουν ακόμη τρία χρόνια μέχρι να δούμε τι πρέπει να γίνει και χρειάζεται ακόμη πολλή δουλειά. Η Ένωση πρέπει να είναι έτοιμη να ανταποκριθεί στα αυξανόμενα και συνεχώς καινούργια εγκλήματα και απειλές και άρα πρέπει επιγόντως να προγραμματίσει την αντιπόκρισή της. Σας ευχαριστώ πολύ και απορροσμένο προσβλέπω στις απορίες σας. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, τώρα προχωράμε στην εισηγήτρια την κυρία Μπορσελίνο και ε, αυτή θα ανοίξει και τη συζήτηση για όσους από τους ευρωβουλευτές θέλουν να παρέμβουν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο της Κόζη για την παρουσίαση την οποία θεώρησα πολύ ενδιαφέρουσα. Χαιρετίζω και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που στην έκθεσή της κατέστησε συγκεκριμένη την προσέγγιση την οποία τα κράτη-μέλη πρέπει να υιοθετήσουν το 2012. Νομίζω ότι ε, υπήρξε μία ε, εκτενής παρουσίαση αλλά πρέπει να λάβουμε υπόψη και το θέμα της εξωτερικής ασφαλείας και νομίζω ότι επ' αυτού πρέπει να εργαστούμε πιο στενά με την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων για να το επιτρέψουμε τύχουμε και θα ήθελα επιπλέον ε, να παρουσιάσω σχετικά ένα κείμενο ε, τον Ιανουάριο το οποίο θα έχω καταρτήσει κατά τη διάρκεια του Δεκεμβρίου ε, θα Ήθελα λοιπόν να υπάρξει ε, μία συγκεκριμένη δράση στους περισσότερους τομείς, τη σοβαρή εγκληματικότητα, την, ε, το κυβέρνο έγκλημα ε, και να τονίσω ότι χρειαζόμαστε συμπληρωματικά μέσα αλλά αυτό το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει πάνω απ' όλα είναι πώς θα αντιμετωπίσουμε το συνολικό πρόβλημα, διότι θεωρώ ότι ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ο ρόλος του δημοκρατικού ελέγχου ουσιαστικά ιδίω για να μπορέσει να προχωρήσει στην εφαρμογή των προγραμμάτων είναι σημαντικός και γι' αυτό το, ο, ο, ο επόμενος κύκλος ο οποίος θα ξεκινήσει το 2013 δεν μπορεί να καθοριστεί χωρίς ε, ε, να συνδυαστεί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και πιστεύω ότι ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι ουσιαστικός και θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη και έναντι της κατανομής των ε, οικονομικών πόρων οι οποίοι θα προβλέπονται στο πολιετές πρόγραμμα. Υπάρχει κι άλλο ένα θέμα επί του οποίου θέλω να σταθώ και αυτό είναι η νομική και δικαστική συνεργασία όπως και η αστυνομική συνεργασία. Πιστεύω λοιπόν ότι έτσι θα επιτύχουμε την ε, ε, εφαρμογή της εσωτερικής στρατηγικής και είναι ένα θέμα που θα τονίσω στην έκθεσή μου διότι η στρατηγική της εσωτερικής ασφαλείας ε, δεν μπορεί να παραβλέψει την εξωτερική διάσταση της ασφαλείας εξού και η Επιτροπή Ελευθεριών εξετάζει το θέμα αυτό συνεργασία με την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων διότι οι ανταλλαγές πληροφοριών διαθεσμικά δεν ικανοποιεί σε αυτό το στάδιο όπως φαίνεται άλλωστε και στα τελευταία ψηφίσματα που υιοθέτησε προσφάτως η Επιτροπή Ελευθεριών ε, σε τομείς όπως η τρομοκρατία και ε, στη την ε, έκθεση Αλφάνο αυτό φάνηκε ε, σαφώς και πέραν της διεκαστικής συνεργασίας θα πρέπει όλοι να συμμετάσχουν εις την εσωτερική πολιτική και να καταρτιστεί ένας δεσμευτικός χάρτης για την δημιουργία ενός χώρου ελευθερίας ασφαλείας και δικαιοσύνης όπου όλα τα θέματα θα είναι άρρηκτα συνδεδεμένα. Είδαμε δηλαδή τι έγινε στο Όσλο εφέτος το καλοκαίρι και το αντιληφθήκαμε διότι γι' αυτό πρέπει να μας απασχολήσει το θέμα των διακρίσεων στα πλαίσια της ασφαλείας και θα πρέπει να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε αποτελεσματικά και ευχαριστώ του συναδέλφους και το Συμβούλιο. Ευχαριστώ. Η κυρία Λάτφορντ έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι η έκθεση αυτή είναι ενδιαφέρουσα. Ίσως ε, τρομάζει κανείς λίγο όταν αντιληφθούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πραγματεύεται τις εσωτερικές υποθέσεις και τη δικαιοσύνη εδώ και 25 χρόνια και ακόμη αντιμετωπίζει σοβαρές προκλήσεις στον τομέα του σοβαρού εγκλήματος και στην ανάπτυξη νέων τομέων που, όπως την αντιμετώπιση του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο. Ε, όσον αφορά το μέγεθος της προκλήσεως του οργανωμένου εγκλήματος πρέπει να παραδεχθούμε ότι ε, είναι τεράστιο και στο έγγραφο αυτό έχουμε πολλές πρωτοβουλίες οι οποίες ανακοινώνονται και νομίζω ότι καλό θα ήταν να δούμε αν τα κράτη-μέλη θα θεωρήσουν, θα σεβαστούν τις υποχρεώσεις οποίες έχουν ήδη αναλάβει διότι έχουμε 8 κράτη-μέλη που δεν έχουν ακόμη κυρώσει την συνθήκη του Συμβουλίου της Ευρώπης για το κυβερνοέγκλημα και αυτό είναι ε, περίεργο ε, δεδομένου στη σημασία που αποδίδει στο κυβερνοέγκλημα ε, οι οι Ηνωμένε Πολιτείες. Ως εκ τούτου βλέπουμε ότι καταρχήν υπάρχουν ήδη ανηλυμένες υποχρεώσεις οι οποίες θα έπρεπε να εφαρμόζονται πλήρω. Προτού ξεκινήσει κανείς νέα νομοθεσία και να καταρτίζει νέες προτάσεις διότι αν υπάρχει ένα σαφές κενό το οποίο πρέπει να καλυφθεί έχει καλός. Αναρωτιέμαι λοιπόν όμως αν δεν θα ήταν καλύτερο να σταθούμε ένα λεπτό και να δούμε αν εφαρμόζονται όλα τα συμπεφωνημένα του παρελθόντος διότι ε, ήδη αυτό είχε γίνει προετών υπό Σουηδική πρωτοβουλία και δεν ξέρω πλέον πού βρισκόμαστε λειτουργικά. Έχω δε την εντύπωση ότι στην Επιτροπή αυτή πολλές φορές σχολιάζουμε τις ανησυχίες μας για πιο μαζική συλλογή στοιχείων ε, για καθενός ε, για τη χρήση ολονών ε, των ηλεκτρονικών μηνυμάτων και ταξιδίων ε, και βλέπουμε ότι εδώ υπάρχει δυστοκία στο να κατασχέσουμε ε, τα περιουσιακά στοιχεία μεγαλοεγκληματίων. Πότε λοιπόν θα βάλουμε κάποια προτεραιότητα στις πράξεις μας διότι βλέπω εδώ στη σελίδα 9 ότι έχει γίνει μεγάλη πρόοδος στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος ιδίω σχετικά με την ομοθεσία των PNR αλλά εφόσον αυτό δεν έχει ακόμη αποφασιστεί θεωρώ ότι είναι μυστηριώδες πως μπορεί να έχουμε προχωρήσει και σε άλλα θέματα που δεν είναι ακόμη υλοποιημένα Πώς είναι δυνατόν να λέμε ότι έχουμε προχωρήσει ε, στην ε, ε, καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Υπάρχουν πολλά στοιχεία, πολλές ιδέες οι οποίες είναι καλές, αλλά πρακτικά κανείς αναρωτιέται πόσο αποτελεσματική έχουμε υπάρξει στην καταπολέμηση αυτή και τέλος μερικά τελευταία θέματα <clears throat> βλέπω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρεται ιδίως στις βίες ακρότητες σε σχέση με την τρομοκρατία και νομίζω ότι καλό θα ήταν να ανταποκριθούν στην έκκληση και να μην μιλούν για τις ριζικές ακραίες μορφές διότι νομίζω ότι δεν θα είναι καλό να μιλάμε, να συσχετίζουμε τους όρους radical και radicalization με τον εξτρεμισμό. Επίσης είδα και μια άλλη ιδέα η οποία έχει υποβληθεί σχετικά με αυτούς οι οποίοι προστατεύουν την προσωπική ζωή, αναφέρεται ιδίω στην ε, προστασία δεδομένων, οι οποίοι ζητούν από τους κατασκευαστές των λογισμικών να εγγυούνται την ασφάλεια των προϊόντων τους, το οποίο βεβαίως δεν πράττουν, διότι ο χρήστης πρέπει να εγγυηθεί. Διότι αν ζητήσουμε εγγυήσεις, τότε ενδέχεται ε, ε, να μην μπορέσουμε να το επιτύχουμε και θα ήθελα αυτό να το συζητήσει η αρμόδια Γενική Διεύθυνση με την υπεύθυνη βιομηχανία. Σας ευχαριστώ. Η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η πρώτη της έκθεση για την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής ε, εσωτερικής ασφάλειας μιλάει στην πρώτη φράση για το δράμα που ζήσαμε στην Ορβηγία όταν ο Άντριος Ράιφεκ σκότωσε πολλούς νέους και ανατείναξε τμήμα ε, και μάλιστα ε, έπληξε ένα ολόκληρο Υπουργείο. Ε, μετά τις πρώτες μελέτες του 2011, οι στατιστικές δείχνουν ότι οι περισσότερες απειλές στην Ευρώπη οφείλονται σε Ισλαμιστικές μονάδες. Είναι η Ισλαμική τρομοκρατία. Είχαμε τις τελευταίες εβδομάδες κάποιες ειδήσει και από τη Γερμανία, όπου ακροδεξιοί τρομοκράτες από την Ανατολική Ευρώπη φαίνεται ότι σκότωσαν πολλούς ε, Τούρκους πολίτες ε, στη Γερμανία και αυτό χαρακτηρίστηκε, αυτή χαρακτηριστεί ως α, ε, α, τουρκικές, α, ε, ως δολοφονίες Τούρκων, αλλά από Τούρκους πολίτες. Αυτή ήταν αρχικά η είδηση που ανακοινώθηκε, αλλά τελικά διαπιστώθηκε ότι η αυτουργία αυτών των δολοφονιών ήταν ε, ακροδεξή και τελικά δεν μπόρεσαν δυστυχώς να εξηχνιαστούν αυτά τα εγκλήματα. Γνωρίζουμε με ακρίβεια ποιες είναι οι απειλές κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά αυτές οι απειλές, γιατί αν οι στατιστικές δείχνουν ότι θα πρέπει να προστατευτούμε κυρίως από Ισλαμιστές, και αυτά λένε οι στατιστικέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση, να μα τι δείξει ξεκάθαρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στην έκθεση του 2010 τη Europol φαίνεται ότι ε, από τι εννέα ε, υποθέσει που ξεχνιάστηκαν μόνο δύο ή τρει ήταν ε, από Ισλαμιστέ. Δεν είμαι εμπειρογνώμων βέβαια, αλλά προ τι να δαπανούμε χρόνο, ενέργεια και χρήμα σε απειλές που δεν είναι σίγουρο ότι γνωρίζουμε την προέλευσή τους έχουμε καταρχήν ως βάση πληροφορίες ε, που δεν είναι πάντα έγκυρες και ακριβείς, γιατί δεν φαίνεται ότι ελέγχονται. Δεν έχουμε σαφή ιδέα για το από πού προέρχονται αυτές οι απειλές. Και είδαμε ότι οι ε, περσινές απειλές δεν είχαν καθόλου ισλαμική, ισλαμιστική προέλευση. Ήταν ε, τελείως διαφορετική φύση. Οπότε αυτή την άποψη πώς είναι δυνατόν να συμφωνήσουμε με τις προτάσεις. Επιπλέον, είναι προβληματική ένταξη του ελέγχου των συνόρων στη στρατηγική ασφάλεια. Γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι που διέρχονται από τα εξωτερικά σύνορα είναι μετανάστες, είναι τουρίστες, είναι άνθρωποι που πολύ ευχαρίστω υποδεχόμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι κατά ανάγκη όσοι τα σύνορα ε, Και νομίζω ότι είναι σφαλμένο να εντάσσουμε την ε, στρατηγική διαχείριση των συνόρων στην στρατηγική εσωτερική ασφάλεια, γιατί δίνει ασφαλμένο μήνυμα για το πώ αντιμετωπίζουμε τα εξωτερικά σύνορα και τη διέλευσή του. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ένα σημείο της έκθεσης αναφέρει ότι καλεί τα κράτη-μέλη, εθαρρύνει μάλλον τα κράτη-μέλη, να συμμετέχουν ενεργώς σε διαλόγους ε, για τη μετανάστευση και την κινητικότητα ε, με την Αφρική και τη Μέση Ανατολή. Σίγουρα θα πρέπει να θαρρύνουμε τα κράτη-μέλη να έχουν τέτοια διάλογο. Γιατί όμως μόνο υπό το πρίσμα της ασφάλειας, καλύτερα υπό το πρίσμα της ε, εμπέδωσης της δημοκρατίας. Νομίζω ότι αν αλλάξουμε αυτή την ε, οπτική γωνία θα δώσουμε ένα καλύτερο χαρακτήρα, γιατί ε, οι επαφές με, τη, με τους γειτονές είναι θέμα συνεργασίας και όχι κατά ανάγκη ζήτημα στρατηγικής εσωτερικής ασφάλειας. Ερωτώ λοιπόν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συμφωνείτε ότι χρειαζόμαστε περισσότερε αποδείξει και τεκμήρια από ανεξάρτητους ελεκτές πριν να καταλήξουμε σε αυθαίρετα συμπεράσματα για τις πηγές της τρομοκρατίας και κυρίως για τις διασυνδέσεις τρομοκρατίας και εργανομένου εγκλήματο. Επίσης χρειαζόμαστε πιο αδιάστατα επιχειρήματα για την πρόταση συρρήκνωση ε, των δαπανών, μια και έχουμε ε, λιγότερη ασφάλεια και μάλιστα σε περίπτωση χρηματοπιστωτικής χρήσης. Απ' την άλλη έχουμε τεράστια και πανηρά προγράμματα όπως το PNR, όπως το πακέτο για τα ΕΦΗ e σύνορα, προκειμένου να ελέγχουμε όλους τους ε, ταξιδιώτες εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προς τι όλες αυτές οι δαπάνες εν μέσω χρηματοπιστωτικής κρίσης. Έχουμε πραγματικά βάσιμο επιχείρημα ότι όλες αυτές οι προσπάθειες αξίζουν τα κονδύλια που τους αφιερώνουμε. Και τέλος, υπέβαλα ερώτηση για την εντολή της Europol. Και από ό,τι κατάλαβα, κανείς δεν μπορεί να το ελέγξει και δεν υπάρχει καν δημοκρατικός έλεγχος της Europol. Παρ' όλα αυτά, στηριζόμαστε στη Europol για όλες μας τις αναλύσεις. Και τελευταία ερώτηση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε ε, με ένα ρόλο στο κέντρο για την ακτίμηση της εσωτερικής ασφάλειας. Ποιος όμως θα λογοδοτήσει, ποιος θα είναι υπόλογος για το κέντρο αυτό και από πού λαμβάνει το κέντρο τις πληροφορίες τις οποίες στηρίζεται. Και τέλος, αν μιλούμε για εσωτερική ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει πρώτα να καταλήξουμε σε έναν ορισμό για το τι είναι εσωτερική ασφάλεια. Γιατί το να αναμειγνύουμε ε, θεομηνίες, τρομοκρατία και οργανωμένο έγκλημα δεν νομίζω ότι βοηθάει σε μια διαφανή αντίληψη της κατάστασης. Ευχαριστώ κυρία Τσίπελ. Just, just let me remind you that... Αλλά να σας υπενθυμίσω ότι ήδη από την αρχή της απογευματινής συνεδρίασης ο κύριος Κουμανέκ με ενημέρωσε ότι κανονικά ε, θα φύγει σε λίγο. Έχει αεροπλάνο ο άνθρωπος. Οπότε επικεντρωθείτε συγκεκριμένε ερωτήσει προς τον κύριο Κουμάνα. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ρωτήσω ή μάλλον να κάνω μία παρατήρηση σε τρία θέματα. Το πρώτο είναι η καταπολέμηση των συνθετικών ναρκωτικών. Ε, υπάρχουν στα κράτη-μέλη οι ίδιες νομοθεσίες για την καταπολέμηση παρανόμων ε, ναρκωτικών και συνθετικών ναρκωτικών ή υπάρχουν διαφορές. Και όσον αφορά τα συνθετικά ναρκωτικά πόσο αποτελεί το διαδίκτυο κλασικό, κλασική οδό εμπορίας έχει ληφθεί υπόψη επίσης θα ήθελα να ξέρω όσο αναφορά την διακίνηση ατόμων κατά πόσο να αναφέρεται κανείς μόνο ε, εις τις δικαστικές σκοπιές και αν λαμβάνεται υπόψη και το θέμα της απασχόλησης και μετά ε, λέχθη ότι ε, το θέμα του κυβερνοεγκλήματος είναι μια πολύ ευρία έννοια για ορισμένους είναι μόνο ε, η εγκληματικότητα στο διαδίκτυο ενώ υπάρχουν και υποκλοπές ταυτότητος. Θα ήθελα να ξέρω καταρχήν εάν δεν θα έπρεπε να μπορέσουμε να ξεκαθαρίσουμε αν χρειαζόμαστε όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία ζητάμε διότι μπορεί να υπάρχει και εκμετάλλευση των στοιχείων αυτών. Μήπως ε, ορισμένα από αυτά τα στοιχεία τα οποία συλλέγονται ε, για να καταπολεμήσουμε την εγκληματικότητα δεν μπορούν ε, να επιτευχθούν με ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση αναβάθμιση του προσωπικού ορισμένων οργανισμών και όσο αναφορά τα ναρκωτικά πόσο μπορεί κανείς να είναι βέβαιος ότι υπάρχει μία ενημέρωση σχετικά με την προστασία χωρίς να χρειάζεται κανείς να περιμένει. Ο κύριος Άλμπρεχτ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θα είμαι πολύ σύντομος γιατί εγώ αναφέρομαι σε ένα θέμα μόνο στην cyber security και cyber crime κυβερνοέγκλημα και ε, ε, ε, ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Ιδίω όσον αφορά το κυβερνοέγκλημα αναφέρομαι στην παιδική πορνογραφία και την πνευματική, κατα, παραβίαση της πνευματικής ιδιοκτησίας και μου φαίνεται αστείο ότι αυτά είναι τα δύο μόνα παραδείγματα τα οποία αναφέρονται και αν, ε, θέλω, εάν συγκεντρώνει κανείς τα δύο θέματα αυτά και τα συνοψίζει σε μία φράση το θεωρώ επίσης περίεργο γιατί ε, το ένα θέμα ε, είναι αυστηρό έγκλημα το οποίο θέλουμε να παρακολουθούμε ιδίως μέσω του διαδικτύου και από την άλλη πλευρά στις περισσότερες περιπτώσεις ε, δεν πρόκειται καν για αδίκημα πρόκειται για ένα παράπτωμα ναι με αξιόπινη πράξη αλλά δεν είναι έγκλημα δεν ανήκει στην ίδια κατηγορία και δεύτερον δεν αντιλαμβάνομαι γιατί σε ένα έγγραφο για την εσωτερική ασφάλεια ε, αναφερόμαστε σε την παραβίαση της πνευματικής ιδιοκτησίας. Θέλουμε καλύτερη επόπτευση του διαδικτύου αλλά εδώ δεν μπορούμε να μπερδεύουμε ε, τα προσωπικά δεδομένα με άλλα θέματα και ε, για, με ε, επιχειρήσεις οι οποίες πουλούν τα προγράμματά τους μέσω του διαδικτύου. Εδώ μιλάμε για ασφάλεια και παραβίαση της πνευματικής ιδιοκτησίας. Τουλάχιστον εγώ έτσι το θεωρούσα. Το θέμα της ανταλλαγής μουσικής και ε, ε, της ε, παραποίησεως δεν με απασχολεί τόσο πολύ εδώ. Η κυρία... Μάλιστα κύριε Πρόεδρε, τρία θέματα. Πρώτον συμφωνώ απόλυτα με αυτά που είπε ο Γιάννο Όλμπρεχτ. Ποιος είναι ο ορισμός της εσωτερικής ασφαλείας. Εκείνος μίλησε για πνευματικά δικαιώματα, διεθνή πνευματικά δικαιώματα η Κομισιόν, μίλησε για απειλέ κατά των πνευματικών δικαιωμάτων. Τι, τι, τι γλώσσα είναι αυτή εννοεί. Και αν καλύπτεται αυτό, τι θα γίνει με την οικιακή βία που δημιουργεί εκατοντάδες θύματα το χρόνο. Γιατί δεν είναι και αυτό απειλή κατά της εσωτερικής ασφαλείας. Πρώτο θέμα λοιπόν ο ορισμός. Δεύτερο θέμα. Η δημοκρατική επιτήρηση. Εδώ υπάρχει ένα τεράστιο έλλειμμα. Γιατί ως εκπρόσωποι των λαών υποχρεωνόμαστε να περνάμε νομοθεσία που μερικές φορές αποφεύγει να βλέπει τα πραγματικά προβλήματα και δεν μπορούμε να ε, τεκμηριώσουμε κατά πόσον αυτά που μας λένε είναι σωστά. Πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη απλώς στο Συμβούλιο και την Κομισιόν ότι όλα αυτά είναι τελείως απαραίτητα, αλλά δεν μπορούμε να το επαληθεύσουμε. Χρειαζόμαστε λοιπόν μηχανισμούς επαλήθευσης. Και τρίτον, αυτό που με εντυπωσιάζει πάντοτε είναι ότι για δέκα και παραπάνω χρόνια ψηφίζουμε ένα μέτρο μετά το άλλο και κάθε φορά που γίνεται κάτι καινούργιο λαμβάνουμε καινούρια μέτρα. Κάτι όμως λείπει πάντοτε, η συνεργασία και η ανταλλαγή απόψεων και πληροφοριών. Κάθε φορά φαίνεται ότι η πληροφόρηση που χρειαζόταν οι διοκτικές αρχές υπήρχε αλλά δεν είχε διατεθεί, είχε παρερμηνευτεί, δεν είχε αναλυθεί σωστά δεν υπήρχε συνεργασία τελικά μεταξύ των διαφόρων υπηρεσιών, χωρών. Κάθε φορά που γίνεται κάτι το διαπιστώνουμε εκ νέου. Γιατί δεν προσπαθούμε να πετύχουμε καλύτερη συνεργασία των υπαρχουσών υπηρεσιών αντί να ψηφίζουμε καινούργιους νόμους. Δεν πρόκειται αυτό να αυξήσει την ασφάλεια. Πάνω απ' όλα χρειάζεται καλύτερη πληροφόρηση και συνεργασία. Εγώ νομίζω και πάντα νόμιζα ότι είναι πικρή ηρωνία το γεγονός ότι οι εγκληματίες συνεργάζονται διαμεθοριακά χωρίς πρόβλημα και υποφελούνται από το άνοιγμα της Ευρώπης. Γιατί δεν συνεργάζονται και οι τίμοι άνθρωποι λοιπόν. Ευχαριστώ. Ο κύριος Φως. Ευχαριστώ. Οι τρεις προλαλήσαντες έχουν ήδη καλύψει πολλά από τα θέματα τα οποία θα ήθελα να ρωτήσω και γι' αυτό θα κάνω σύντομες περαιτέρω ερωτήσεις. Η αναγνώριση ότι η παράνομη ε, μετακίνηση υπάρχει εξ Ανατολών της Γερμανίας ε, είναι αποδεδειγμένη διότι νομίζω ότι εντωμεταξύ η παράνομη μετακίνηση και μετανάστευση έρχεται από τις δυτικές χώρες. Επίσης ε, εδώ νομίζω ότι ε, πρέπει να ε, ε, συνδεθούμε περισσότερο σε δίκτυο για την προστασία των δεδομένων για να υπάρχει μεγαλύτερη ασφάλεια ή αυτά τα θέματα δεν εξετάζονται ακόμη. Ευχαριστώ. Ακούσαμε για τα προγράμματα και ιδίως ε, και για πολιετή προγράμματα και είπατε ότι η κόζη δεν ενδιαφέρεται με να λαμβάνει λειτουργικές αποφάσεις ή να νομοθετεί αλλά βεβαίως η κόζη δεν είναι αστυνομία και δεν μπορεί να λάβει λειτουργικές αποφάσεις παρόλο που ορισμένες αποφάσεις ή ορισμένα είδη αποφάσεων θα έπρεπε να αναλαμβάνονται. Το δεύτερο είναι σωστό ότι η κόζη δεν είναι νομοθετικό όργανο άρα δεν μπορεί να νομοθετήσει αλλά φαντάζομαι όπως ανέφερε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι ορισμένοι εμπνέονται από την, ε, εργασία σας. Αν αυτό δεν ευσταθεί ε, θα ήθελα να ξέρω ε, ποια είναι η μεγαλύτερη, πιο αποτελεσματική επιχείρηση η οποία έχει αναλυφθεί η οποία οφείλεται εις την κόζη. Δηλαδή κατά πόσον η κόζη έχει συμβάλει στην ασφάλεια όλων μας. Επαναρχόμαστε τώρα ε, στον εκπρόσωπο της Κόζη τον κύριο Κουμάνη και στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κύριο Ελμέιντα. Ε, κύριε Κουμάνη, θα λάβετε εσείς πρώτο το λόγο, ώστε να προλάβετε και την πτήση σας μετά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ξεκινήσω με την τελευταία παρέμβαση. Φυσικά, η Επιτροπή Κόζη για πρώτη φορά εφαρμόζει αυτό τον ε, ευρωπαϊκό κύκλο πολιτικής. Και μάλιστα βρισκόμαστε σε μια πολύ κρίσιμη φάση όπου καθορίζουμε τους στρατηγικούς ε, στόχους και τώρα εκπονούμε τα επιχειρησιακά σχέδια δράσης. Αυτά τα σχέδια δράσης, όπως είπα και προηγουμένως στην παρουσίασή μου, θα αρχίσουν να εφαρμόζονται από τον Ιανουάριο και μετά. Βέβαια τα επιχειρησιακά σχέδια δράσης είναι πολύ χρήσιμα εργαλεία και θα χρησιμοποιηθούν και στις επιχειρήσεις που θα, θα προγραμματιστούν και η προσέγγιση αυτή έχει πολλά θετικά προγνωστικά και είναι ελπιδοφόρα αλλά Βρισκόμαστε σε μια διαδικασία να το γίγνεσθε και δεν ξέρουμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Είναι τόσο αίσιο όσο περιμένουμε. Είναι μια διαδικασία που μόλις πρόσφατα ξεκίνησε και μαθαίνουμε στην πορεία. Εγώ ευελπιστώ ότι στο μέλλον θα μπορέσουμε να σας δώσουμε και πιο διεξοδικές και πιο απτές πληροφορίες για τις επιτυχίες αυτού του μηχανισμού μετά την πρώτη χρονιά εφαρμογής των επιχειρησιακών σχεδίων δράσης. Σας ευχαριστούμε κύριε Κουμάνεκ, ο κύριος Νούνης Δελμέιντα. Από... Στο, στο μέτρο που η στρατηγική αυτή καλύπτει το σύνολο της πολιτικής εσωτερικής ασφάλειας και υπερβαίνει τις ε, δικές μου στενές αρμοδιότητες, δεν είμαι βέβαια, ότι θα καταφέρω να απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις. Θα σας ε, δώσω πάντως ε, κάποια στοιχεία. Η κυρία Λάντφορντ είπε ότι θα πρέπει να επανεφεύρουμε τον τροχό, θα πρέπει να ξεκινήσουμε από αυτό που υπάρχει, να το αναπτύξουμε και να το αξιοποιήσουμε. Και σε μεγάλο βαθμό αυτό κάνουμε. Όχι μόνο αυτό όμως, γιατί υπάρχουν όντως και καινοτόμες πρωτοβουλίες. Αλλά δεν ευσταθεί ότι αδιαφορούμε πλήρω για τα υφιστάμενα και, τους, και δεν αξιοποιούμε τα ήδη υπάρχοντα. Ίσα ίσα τα αξιοποιούμε και όλο και περισσότερο και το 2012 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προβεί σε μια ενδελεχή αξιολόγηση και θα υποβάλει συστάσεις για τη βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των αστυνομικών δυνάμεων. Και μάλιστα θα δούμε πώς έχουν λειτουργήσει η Σουηδική Πρωτοβουλία και η Συμφωνία της ΠΡΟΥΜ χάρη σε μια ενδελεχή αξιολόγηση που θα γίνει μετά από το πρώτο έτος εφαρμογής. Θα διαμορφώσουμε και τη στρατηγική μας για την εκπαίδευση και την κατάρτιση των αστυνομικών δυνάμεων. Θα δούμε ποια είναι η καλύτερη εκπαίδευση προκειμένου να βελτιωθούν τα εφόδια των αστυνομικών δυνάμεων τώρα που δρούν πλέον σε ένα πανευρωπαϊκό πλαίσιο. Δεν πρόκειται να επανεφεύρουμε ούτε μέτρα καινούργια ούτε καινούριου θεσμού, αλλά θα χρησιμοποιήσουμε τους υπάρχοντες θεσμούς ε, τις τελευταίες 15 ετίες και θα τους ενισχύσουμε, θα τους αξιοποιήσουμε. Επίσης, οι οργανισμοί Europol και CIPOL ε, θα υποστούν μια αξιολόγηση για να δούμε με, μέχρι στιγμής πώς λειτουργήσαν. Διαφωνώ με την κυρία Σαρτζεντίνη που είπε ότι η Europol εκφεύγει του κοινοβουλευτικού ελέγχου ότι έχει ένα είδος χέρι ενός είδους λάθος. Υπόκειται στον κοινοβουλευτικό έλεγχο και η Europol και θα υποβάλουμε και σχετικά μέτρα, αλλά ήδη ο προπολογισμό της Europol υπόκειται στην έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ο, ο υπολογισμό είναι πολύ ισχυρό εργαλείο για έλεγχο. Και φαντάζομαι και η Europol και τα τα διοικητικά της όργανα. Πολύ ευχαρίστω ε, θα υποστούν τον έλεγχο και της δικής σας επιτροπής και πολύ ευχαρίστω θα λογοδοτήσουν για τις δράσεις που αναλαμβάνουν. Δεν νομίζω ότι είναι σωστή, σωστός αυτός ο χαρακτηρισμός της Europol ως οργανισμού που εκφεύγει του κοινοβουλευτικού ελέγχου ή είναι υπεράνω τέτοιου ελέγχου. Η κυρία Λάτφορντ έκανε και ένα ηρωνικό σχόλιο για το PNR και το πακέτο πάταξης της διαφθοράς και ότι δεν έχει αντιμετωπιστεί κάποιο συγκεκριμένο οργανωμένο έγκλημα. Μέχρι στιγμής υποβάλλουμε προτάσεις και ελπίζουμε κάποια στιγμή να υλοποιηθούν ώστε όντως να καταφέρουμε να πατάξουμε και εμπράκτος το οργανωμένο έγκλημα. Αλλά δεν μπορούμε να περάσουμε στην πράξη αν δεν έχουμε προηγουμένως τις προτάσεις, ε, δεν έχουμε διαμορφώσει την πολιτική και δεν έχουμε θεσπίσει κάποια μέτρα. Δεν είναι σωστό να λέμε ότι με την πρωτοβουλία για το οποίο είναι το πακέτο κατά της διαφθοράς δεν καταφέρουμε να καταπολεμήσουμε και το οργανωμένο έγκλημα. Η κυρία Σαρτζεντίνη είπε ότι δεν θα πρέπει να εντάσσουμε τη διαχείριση των συνόρων ή τα σύνορα στους μηχανισμούς εσωτερικής ασφάλειας. Εδώ μιλούμε όμως για μια στρατηγική εσωτερικής ασφάλειας και είπαμε ότι στα πλαίσια αυτή τη στρατηγική εσωτερική ασφάλεια και τα σύνορα θα μπορούσαν να, χρησιμοποιήσουν, να χρησιμοποιηθούν ω εργαλείο για την καταπολέμηση τη τρομοκρατία και του οργανωμένου εγκλήματο. Αυτό δεν σημαίνει ότι η αποκλειστική χρησιμοποίηση των συνόρων είναι για την καταπολέμηση τη τρομοκρατία και του οργανωμένου εγκλήματο. Απλώ εντάσσονται και αυτά στην στρατηγική. Αυτό περιλαμβάνει το άγγραφο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η κυρία Τσίπελ είπε ότι η καταπολέμηση του, των παράνομων ενεργειών θα πρέπει να, να περιλαμβάνει και ε, λαθρεμπόριο οποιασδήποτε μορφής. Αλλά εγώ δεν είμαι αρμόδιος για αυτά τα θέματα οπότε δεν μπορώ να το σχολιάσω. Ό,τι αφορά την προστασία των δεδομένων, από ό,τι ξέρετε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, θα προτείνει αναθεώρηση της σχετικής νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων. Η πρόταση αυτή θα είναι έτοιμη προς το τέλη του έτους και σε αρχές του επόμενου έτους προκειμένου να τροποποιηθεί το ισχύον πλαίσιο για την προστασία των δεδομένων. Η κυρία Ιντβελτ είπε ότι θα πρέπει και η ενδοοικογενειακή βία να θεωρηθεί ως ε, συγκεκριμένη και πολύ σοβαρή μορφή εγκλήματος στον κυβερνοχώρο. Δεν είμαι κατά και φαντάζομαι ότι οι αρμόδιοι για το θέμα αυτό συνάδελφοι δεν θα διαφωνήσουν με την κυρία Ίντφελτ. Διαφωνώ πάντως με την εκτίμησή σας ε, ότι δεν διαπιστώθηκε ε, ανάγκη κάποιων μέτρων που παρεμβαίνουν στην ιδιωτική σφαίρα, όπως είναι ορισμένα τα μέτρα του PNR. Διαφωνώ. Είχαμε συζήτηση και στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών και είχαμε αυτά παραδείγματα που κατέδειξαν την ανάγκη ε, της χρήσης του PNR προκειμένου να διαλευκανθούν ε, συγκεκριμένα εγκλήματα και να διεκπαιρεωθούν ε, έρευνες. Και πολλές φορές ε, διαπιστώθηκε η ανάγκη του PNR στην διαλεύκανση συγκεκριμένων εγκλημάτων και στην πάταξη κάποιων τρομοκρατικών ενεργειών. Ο κύριος Αξελβός ρώτησε αν ε, αναλύουμε κάποια μέτρα για στοιχεία επιβατών. Ναι, έχουμε ήδη καταθέσει πρώτη μια οδηγία για μια ευρωπαϊκή πρόταση σε ό,τι αφορά τα δεδομένα των επιβατών. Και προς το παρόν δεν έχω να προσθέσω τίποτε άλλο. Λυπούμε αν εκνεύρισα μερικούς ή απογοήτευσα κάποιους ευρωβουλευτές ε, ε, γιατί δεν απάντησα στις ερωτήσεις τους, αλλά πολύ ευχαρίστω θα διαβιβάσω τις ερωτήσεις στους αρμόδιους συναδέλφους που είναι πιο κατάλληλα προετοιμασμένοι και κατατοπισμένοι για να δώσουν σχετικές απαντήσεις. Σας ευχαριστούμε και σας κύριε Αλμέιδα και τον κύριο Κουμάνεκ. Αυτά προς το παρόν. Νομίζω ότι συγκεντρώσαμε αρκετό υλικό για τη δική μας έκθεση ίδια πρωτοβουλία. Ε, στην οποία η συγκήτρια είναι η κυρία Μπορσελίνο. Και αν δεν υπάρχουν άλλα σχόλια, μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Ε, αποχαιρετώντας τον κύριο Κουμάνε και ευχαριστώντας τον για τη συμμετοχή στη συζήτηση. Σας ευχαριστούμε και θα τα πούμε άλλη φορά. Και με τήρηση του χρονοδιαγράμματός μας μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο σημείο. Εμείς είμαστε πραγματικά συνεπείς στο χρόνο μας, αλλά δεν έχει έρθει ακόμη ο εισηγητής μας, ο κύριος Μωράες. Το σημείο 10 αφορά την έκθεση Μωράες για τον κανονισμό του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου σχετικά με τη θέσπιση ενός μηχανισμού αξιολόγησης και παρακολούθησης ε, για, την, ε, για, την, για τους εποχιακούς εργαζόμενους. Α, στο μεταξύ κατέφθασε και ο εισηγητής μας, ο κύριος Κλοντ ή δεν έχει έρθει ακόμη. Μπορούμε να τον καλέσουμε παρακαλώ. Να του δώσουμε μια ευκαιρία να εμφανιστεί. Είναι στο δρόμο ο κύριος Μωράες. Τον περιμένουμε να πάσα στιγμή. The Subject. As I tell you, we got a discussion to go on seasonal workers. Επαναλαμβάνω, θα εξετάσουμε Τη προποθέσει όδου και διαμονή υπηκόων τρίτο χωρών με σκοπό την εποχιακή απασχόληση. Ο κύριο Μωράε υπέβαλε το σχέδιο έκθεσή του την Άνοιξη. Η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών είχε οριστεί πριν τι θερινέ διακοπέ. και έκτοτε ο κύριο Μωράε συνέχισε την επεξεργασία τη έκθεση με του κοιόδη ηγητέ στην Επιτροπή Απασχόληση, προκειμένου να καταλήξει συμβιβαστικέ τροπολογίε. Θα θυμάστε ότι έχουμε εδώ εφαρμογή του άρθρου 50, συνεργασία με την Επιτροπή Απασχόληση. Με το που θα καταθέσει ο κ. Μωράη, θα μα κάνει την παρουσίαση τη έκθεσή του, αλλά στο μεταξύ μπορούμε να ακούσουμε τον εκπρόσωπο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, του Συμβουλίου συγγνώμη, για να μας ενημερώσει για τις εξελίξεις και κατόπιν να ακούσουμε και τον κύριο Κοφεράτη που είναι ο εισηγητής της Επιτροπής Απασχόλησης για το ίδιο θέμα. Ας περιμένουμε λίγο ακόμα όμως τον κύριο Μωράες. Calling off a break. Let's wait for Mr. Moraes for a minute. Προτιμώ να μην διακόψουμε. Θα περιμένουμε κανένα λεπτό μέχρι να έρθει ο κύριος Μωράες.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 Καλησπέρα κύριε Μωράες, και καλώς ήρθατε. Η απουσία σας, η παρουσία σας, η αναμονή της παρουσίας σας α, ε, α, ε, δημιούργησε υψηλότερες προσδοκίες. Σας περιμένουμε πώς και πώς για να μας παρουσιάσετε την έκθεσή σας για τους εποχικά απασχολούμενους. Μετά θα ακούσουμε την Πολωνική Προεδρία, τον εκπρόσωπο του Συμβουλίου και μετά τον κύριο Κομφεράτη, τον εισηγητή της Επιτροπής Απασχόλησης για να δούμε πώς έχουν τα πράγματα και στην Επιτροπή Απασχόληση. Πρώτα όμως, αν το επιθυμείτε, έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, με συγχωρείτε που καθυστέρησα αλλά δεν αισθανόμουν καλά και πήγα στην ιατρική υπηρεσία. Δεν αισθανόμουν πολύ καλά, πράγμα το οποίο δεν είναι συνηθισμένο για μένα και ζητώ συγγνώμη από όσους με περίμεναν. Αγαπητοί συνάδελφοι, ε, έγινε σήμερα μία πολύ σημαντική συνεδρίαση μεταξύ σκιωδών εισηγητών και ε, προσωπικού και πρέπει να πούμε ότι όλοι έχουν δουλέψει σκληρά για την κατάρτιση του φακέλου και αυτό που θα σας πω ουσιαστικά αναφέρεται ε, στο αποτέλεσμα της συνεργασίας όλων των σκιωδών διότι αυτό το θέμα των εποχιακών εργαζομένων είναι πολύ σημαντικό και έχει γίνει πολλή δουλειά και στις άλλες ομάδες για να φτάσουμε στη σημερινή κατάσταση. Θα ήθελα λοιπόν καταρχήν να σας πω ότι ουσιαστικά αναφερόμαστε στη συμβιβαστική πρόταση της ε, ε, ε, Τροπής Ελευθεριών διότι υπήρξε μία αποδοχή πολύ θετική για την Επιτροπή και θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή της Επιτροπής Απασχόλησης τον κύριο Κοφεράτη ο οποίος είναι εδώ σήμερα και θα μας πει πώς ε, κατέληξε η ψηφοφορία της περασμένης εβδομάδας σχετικά με τους εποχιακούς εργαζομένους αλλά προς στιγμή θα ασχοληθούμε μόνο με τις αρμοδιότητες της Επιτροπής μας Ελευθεριών και πρέπει να πω ότι υπήρξε συμφωνία σε όλα τα βασικά θέματα και ε, στο τέλος φτάσαμε τα ένα ή δύο θέματα όπου υπήρχε ακόμη συζήτηση όσον αφορά τους τομείς ε, και τις ε, ρυθμίσεις. Από όταν ανέλαβα αυτή την έκθεση πρέπει να πω ότι όλα τα θέματα έχουν καταλήξει σε μία κοινή διεκπαιρέωση και σε συμβιβαστικές τροπολογίες. Υπήρξε και το θέμα της ε, διαβουλεύσεως με τους κοινωνικούς εταίρους που ήταν σημαντική και που με βοήθησε ο κύριος Κοφεράτη και οι σκιώδεις συνεργάστηκαν για να καταλήξουμε σε μία καλή λύση επί του θέματος και να δούμε ε, πώς θα το επιτύχουμε ε, και πώς οι κοινωνικοί εταίροι θα εμπλακούν. Όσον αφορά το θέμα αυτό λοιπόν είδαμε ότι εξετάσαμε και το θέμα της κατοικίας και των ρυθμίσεων που απαιτούν αυτοί οι εποχιακοί εργαζόμενοι και νομίζω ότι και πάλι η ρύθμιση ήταν ικανοποιητική. Πρόκειται για περιορισμένη διάρκεια παραμονής 6 έως 12 μηνών, αλλά αντιλαμβανόμαστε ότι τα κράτη-μέλη ζητούν να υπάρξει μία περίοδος 5 έως 9 μηνών ε, και θα θέλαμε τα κράτη να έχουν κάποια ευελιξία για να επιλέξουν τον χρόνο που τους, της επιλογής τους ε, μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Για την προστασία των εποχιακών εργαζομένων όλοι οι σκιώδεις ε, τόνισαν ε, την προστασία του νομικού συστήματος, του συστήματος παραπόνων χωρίς να έχουμε υπερβολή πολιτικό γραφειοκρατικό φόρτο. Και τέλος τα δύο σημεία τα οποία νομίζω ότι ακόμη χρειάζονται επεξεργασία είναι καταρχήν η εμβέλεια και δεύτερον τα κριτήρια επιλογής στα δύο αυτά θέματα που είναι πολύ περίπλοκα για την ε, Επιτροπή ΛΥΜΠΕ νομίζω ότι θα υπάρξουν διαφορές διότι καταρχήν όσον αφορά ε, το στόχο που επιζητεί αυτή η ρύθμιση δηλαδή εάν πρόκειται ε, ε, για πολίτες οι οποίοι έρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους από οποιαδήποτε άλλη κατηγορία θα πρέπει να διαπιστώσουμε ότι υπάρχουν διαφορές και οι σκιώδεις προσπαθούν να τις επιλύσουν αλλά σέβομαι όλες τις αποφάσεις που έχουν διατυπωθεί επί του θέματος αυτού και είμαι στη διάθεσή σας σχετικά με την εμβέλεια αυτή. Επίσης αναφορά τα κριτήρια επιλογής. Δεν εξετάσαμε ε, μόνο τα άρθρα αλλά ε, επίσης ε, και άλλα για πολύ προσεκτικά για να μην δώσουμε λανθασμένο μήνυμα σχετικά με την είσοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θέλαμε να υπάρξει ε, ε, σύγχυση με άλλα πολιτικά μηνύματα. Πρέπει λοιπόν να λύσουμε τις δύο αυτές συμβιβαστικές λύσεις που συνεχίζουν να είναι περίπλοκες και ελπίζω ότι μέχρι τον Ιανουάριο που θα ψηφίσει η Επιτροπή θα έχουν επιληθεί και τα δύο αυτά τελευταία θέματα. Τέλος πρέπει να σας πω ότι η ε, οι σκιώδεις με βοήθησαν να παρουσιαστούν πολλά θέματα και θα ήθελα να ακούσω και την άποψη του Συμβουλίου επί αυτού. Σας ευχαριστώ. Τώρα η Πολωνική Προεδρία, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ θερμά τον εισηγητή για την στενή συνεργασία που έχουμε στα πλαίσια του θέματος αυτού. Το θέμα και έκθεση είναι πολύ σημαντική γιατί έχουμε μόνιμη ενημέρωση και ανταλλαγή πληροφοριών ε, μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου και αυτό είναι χρήσιμο. Σε ό,τι αφορά για την εξέλιξη των εργασιών, μέχρι στιγμή είχαμε τρει ε, συσκέψει ε, και συναντήσει σε ό,τι αφορά την οδηγία για του εποχιακά εργαζομένου. και στι 2 Δεκεμβρίου θα έχουμε την τελευταία αυτή συνάντηση και θα έχουμε και την συνεδρίαση της ειδική ομάδας εργασίας που ασχολείται με το θέμα αυτό. Σε ό,τι αφορά τη διεξαγωγή των εργασιών, στην τελευταία ε, συνεδρίες στο Συμβούλιο ασχοληθήκαμε με ειδικά ζητήματα που αφορούν τις ε, θεωρήσεις και την ε, βραχία και μέση διάρκειας διαμονή. Είχαμε τη διαμονή μέχρι τριών μηνών και διαμονή μεγαλύτερης διάρκειας, γιατί έχουμε δύο διαφορετικά καθεστώτα που διέπουν αυτές τις διάρκειες και είναι πολύ περίπλοκη η διαφοροποίηση και υπάρχουν φυσικά και κριτήρια υποδοχής ε, ανάλογα με τη διάρκεια των ε, ανθρώπων αυτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα άλλο θέμα που απασχόλησε το Συμβούλιο ήταν κάποια κοινωνικά ζητήματα και συνέπειες αυτής της οδηγίας και μάλιστα η ε, ομάδα εργασία για τα θέματα απασχόλησης και η Επιτροπή Απασχόληση ασχολήθηκαν ιδιαίτερα με το θέμα αυτό. Ένα θέμα που έμεινε εκρεμέ στο Συμβούλιο και ελπίζουμε ότι θα διευθετηθεί την επόμενη, στην επόμενη συνεδρίαση τη Δευτέρα Δεκεμβρίου είναι να καταλήξουμε σε μία συμβαστική λύση για το έγγραφο αυτό και να σας την παρουσιάσουμε, αν όχι κατά το τέλος της ε, Πολωνικής Προεδρίας, τουλάχιστον στις αρχές της επόμενης Προεδρίας. Και μάλιστα θα έχουμε και μια επόμενη συνεδρίαση στι αρχέ Δεκεμβρίου και θα σα ενημερώσουμε διεξοδικά για την πορεία των εργασιών στο Συμβούλιο. Σε ό,τι αφορά τι ερωτήσει του εισηγητού, ό,τι αφορά τη διάρκεια διαμονή για του εποχιακά απασχολούμενου ε, στην επικράτεια των κρατών μελών, η πρόταση του Συμβουλίου είναι 5 με 9 μήνες. Ε, αυτή βρίσκεται επιτάπητος. Είναι συμβαστική πρόταση και προσπαθούμε να πείσουμε τις χώρες ε, που έχουν πολύ μεγαλύτερη διάρκεια διαμονής ε, που εμπίπτει σε αυτό το χαρακτηρισμό της εποχικής απασχόλησης. Πάντως πιστεύω ότι αυτή η ελαστική ρυθμίση που προβλέπουμε, 5 με 9 μήνες, θα μας επιτρέψει να καταλήξουμε σε συμβασμό στο Συμβούλιο. Με ιδιαίτερη ικανοποίηση διαβάσαμε και την τελευταία εκδοχή του, του Κοινοβουλίου που μιλά για διάρκεια 6 με 12 μήνες. Πολύ καλή πρόταση, σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την εκπρόσωπο της Πολωνικής Προεδρίας και τώρα να δώσω το λόγο στον ε, κύριο Κονφεράτη να μας πει πώς ε, διεξήχθη η ψηφοφορία στην Επιτροπή Απασχόλησης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα επί τη ευκαιρία να ευχαριστήσω θερμά όχι μόνο τον Κλοντ Μωρές, αλλά και όλους τους κοιόδης ηγητές της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών. Προσπαθήσαμε από κοινού με τους κοιόδης και στην Επιτροπή σας και στην Επιτροπή Απασχόλησης ε, να συνεργαστούμε στενά. Αυτό βέβαια οδήγησε μια πιο χρονοβόρα ίσως και πιο ε, κοπιαστική διαδικασία, αλλά νομίζω ότι τα αποτελέσματα μπορούν να μας ικανοποιούν όλους και μας κάνουν υπερήφανος. Στην Επιτροπή Απασχόλησης ε, εγκρίναμε με σημαντική πλειοψηφία το κείμενο και αυτό είναι πολύ σημαντικό και το πιο σημαντικό ακόμη για μένα θέμα είναι το γεγονός ότι επί της ουσίας ε, ψηφίσαμε μόνο τις συμβαστικές ε, προτάσεις. Και μάλιστα ήταν πολύ μακροσκελής αυτές οι συμβαστικές προτάσεις, γιατί στη διαμόρφωσή του συμμετείχαν σχεδόν όλες οι πολιτικές ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Καταλήξαμε όμως σε συμβιβασμό και σε πέρας που κατά τη γνώμη μου μπορεί να χαρακτηριστεί αίσιο. Επί της ουσίας, καθορίσαμε και μάλιστα με ακρίβεια τι σημαίνει και τι θα πρέπει να συνιστά ισότιμη μεταχείριση μεταξύ των ε, εποχιακά εργαζομένων που διαμένουν στην Ευρώπη και των εποχιακών εργαζομένων που έρχονται ε, εκτός από τρίτες χώρες και που διαμένουν και εργάζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε τομείς ε, που μας ανέφερε προηγουμένως ο Κλοντ. Ένα άλλο θέμα που επιλύσαμε ήταν ένα μικρό αλλά διόλο αμεληταίο πρόβλημα γιατί υπήρχε ένα κενό εξαιτίας ενός ορίου που υπήρχε στην οδηγία για την απόσπαση των εργαζομένων και τις οδηγίες για τους ε, εποχιακά απασχολούμενους. Στην οδηγία για τους εποχιακά απασχολούμενους αναφερόταν ε, ένα ειδικό ε, ένας ειδικός κατάλογος προϋποθέσεων που ήταν χαρακτηριστικές για τους εποχιακά απασχολούμενους. Ενώ στην οδηγία για τους αποσπασμένους δεν αναφέρονται καν οι εποχιακά απασχολούμενοι. Υπήρχε ένα κενό λοιπόν, γιατί κανένας φυσικά δεν μπορεί να καλύπτεται από δύο οδηγίες και κανένας ε, δεν μπορεί να μένει ακάλυπτος από, πιο, από καμία οδηγία. Μερικές φορές αυτό το κενό, ακόμη και είναι μικρό, δημιουργεί πρόβλημα. Είπαμε λοιπόν με σαφήνεια ότι οι εποχιακά απασχολουμένοι δεν μπορούν να υπόκειται σε απο, αποσπάσεις, ε, να αποσπώνται δηλαδή σε άλλο κρατός μέλος για να παράσχουν εκεί την εργασία τους. Δεν μπορεί να είναι και εποχικά απασχολούμενοι και αποσπασμένοι εργαζόμενοι. Νομίζω ότι η ψηφοφορία διεκπαιρεώθηκε πολύ θετικά και θα ήθελα ένα τελευταίο σχόλιο σε ό,τι αφορά τη διάρκεια τη σύμβαση ενό εποχιακά απασχολούμενη. Με τη συμφωνία όλων των πολιτικών ομάδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επιλέξαμε την εξάμηνη προθεσμία αλλά ο, το εξάμηνο όχι για το διαχειριστικό έτος, αλλά για ένα δωδεκάμηνο μέσα αυτό το δωδεκάμινο θα πρέπει να εντάσσεται αυτή η εξάμηνη διάρκεια. Νομίζω ότι είναι η πιο αποτελεσματική λύση. Εξετάσαμε βέβαια και την πιθανότητα να διαρκεί 5 με 9 μήνες μια εποχή και απασχόληση, αλλά 9 μήνες είναι μεγάλη διάρκεια. Δεν μπορεί να είναι εξορισμού εποχιακή μια απασχόληση που διαρκεί 9 μήνες και ε, υπάρχει αυτό το θέμα του ημερολογιακού έτους, για παράδειγμα. Κάποιος εργαζόμενος που έρχεται για να απασχοληθεί στις χειμερινές διακοπές σε ένα ξενοδοχείο, θα εργαστεί για μερικούς μήνες, που μπορεί να είναι το τέλος ε, ε, του έτους και η αρχή του επόμενου έτους. Μπορεί να εργάζεται από Νοέμβριο με Φεβρουάριο. Δηλαδή, καλύπτει δύο διαφορετικά ημερολογιακά έτη. Ξεπερνά δηλαδή τα όρια ενό έτους. Αυτό όμως σημαίνει ότι η σύμβασή του θα πρέπει να παραταθεί για μεγαλύτερο διάστημα. Νομίζω ότι με το κριτήριο του εξαμήνου που υπολογίζεται όχι με βάση ένα ημερολογιακό έτος, αλλά με βάση ένα δωδεκάμινο. Έτσι καλύπτεται και αυτή η πιθανότητα. Και το 12 μήνο αρχίζει να μετρεί από τη στιγμή έναρξη της ε, διάρκεια τη σύμβαση. Καταλαβαίνω γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιμένει στο 9 μήνο, αλλά είμαι τη γνώμη ότι αν ε, υιοθετήσουμε αυτή την πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που πέρασε με μεγάλη πλειοψηφία στην Επιτροπή Απασχόληση, οι επιφυλάξει που υπάρχουν μέχρι στιγμή στο Συμβούλιο ε, θα μπορούσαν κάλλιστα να έρθουν. Θα ήθελα και πάλι να ευχαριστήσω θερμά όλου όσου συνέβαλαν στη διαμόρφωση αυτού του αποτελέσματος για την πολύ καλή θέληση που έδειξαν και την προθυμία τους για συνεργασία γιατί πραγματικά ήταν λεπτά και δύσκολα τα θέματα και ήταν, θα ήταν πολύ δύσκολο να βρούμε τόσους πολλές συνενετικές λύσεις αν δεν είχαν δείξει αυτόν τον ενθουσιασμό και τη ζέση όλοι οι συμμετέχοντες γιατί χάρη σε αυτό το πάθος και τη ζέση καταλήξαμε σε πολύ θετικές εξελίξεις. Ευχαριστούμε κύριε Κομφεράτη και τώρα Open Room. Η κυρία Σαργεντίνη πρώτη. Ευχαριστώ και σας και τον κύριο Μωράης για τις συμβιβαστικές του τροπολογίες που λάβαμε μόλις σήμερα. Πρώτον, θα ήθελα να πω κάτι για το εύρος. Η πρόταση λέει ότι πρέπει όσοι ζητούν άσυλο να μπορούν ώσπου να βαρθεί απόφαση για την τύχη τους να εργάζονται και οι πράσινοι το δέχονται αυτό αλλά εξαρτάται από το κατά πόσον το κράτος, το κάθε κράτος επιτρέπει στον αιτητή ασύλου να εργάζεται. Εάν ναι, τότε πρέπει να μπορεί να εργαστεί και ως εποχιακός εργαζόμενος. Το θέμα τώρα είναι οι παράνομοι μετανάστες. Αυτοί αν είναι να εκδιωχθούν από μια χώρα με το κεφάλι ψηλά δεν πρέπει και αυτοί να μπορούν να εργάζονται ως εποχιακοί. Αυτό οι πράσινοι το δέχονται γιατί είναι και αυτό ένας τρόπος να φανεί ότι οι παράνομοι μετανάστες πρέπει να έχουν και αυτοί μια εναλλακτική λύση για να μπορούν να επιστρέψουν στη χώρα τους και να καταφέρουν κάτι στη ζωή τους. Η πρόταση οι εποχιακώς εργαζόμενοι να πρέπει να υπογράφουν ένα έγγραφο στην αρχή της σύμβασής τους και να υπόσχονται ή να ορκίζονται ότι θα φύγουν μετά θα καταλήψουν τη χώρα όταν λήξει το συμβόλαιό τους για μας είναι κάτι το υπερβολικό. Αρκεί ότι το συμβόλαιο θα έχει ημερομηνία λήξεως. Δεν χρειάζεται να ορκίζονται και τα προφανή. Εμείς δεν το δεχόμαστε αυτό. Τελευταίο. Ένα ερώτημα προς την Κομισιόν για τις άδειε αντί για θεωρήσεις. Συζητιέται λένε αυτή τη στιγμή στο Συμβούλιο τι ακριβώς χρειάζεται. Αν μπει κανείς σε μια χώρα με μια προσωρινή θεώρηση δεν θα έχει το δικαίωμα εργασίας αφού θα είναι τρίμηνη η θεώρηση ενώ εμείς μιλάμε για εξάμηνη απασχόληση αλλά η άδεια δεν είναι το ίδιο. Θα θέλαμε λοιπόν η Κομισιόν να μας λύσει το νέο αυτό πρόβλημα. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, είναι προφανές ότι οι εποχιακοί δεν πρέπει να πληρώνονται κάτω από τον κατώτερο μισθό ή σε απαράδεκτες συνθήκες. Γιατί μερικές φορές είναι και απάνθρωπες καθαρά οι συνθήκες απασχόλησής τους και έτσι βέβαια υπονομεύουν και την αγορά εργασίας γενικότερα. Αυτά που είδα πριν από 1,5 χρόνο για στους εποχιακούς ήταν τρομακτικά. Λοιπόν, μάθαμε ότι και οι, τοπικός, και οι τοπικοί εργαζόμενοι πέραν των εποχιακών και αυτοί πληρώνονταν κάτω από τον κατώτατο μισθό. Το θέμα παραμένει γιατί απασχολούνται οι εποχιακοί γιατί απασχολούνται εποχιακοί από μακρινές χώρες εφόσον και οι, τοπικός, και οι τοπικοί εργατες έχουν μεγάλη ανεργία. Είναι αποδεκτό να παίρνουν επιδόματα ανεργίας οι τοπικοί ενώ απασχολούνται οι εποχιακοί από άλλες χώρες. Όλοι οι μετανάστες μπορεί να χρειαστεί δυστυχώς να εργαστούν με αυτές τις απαράδεκτες συνθήκες και αυτό διότι και αυτό εξηγεί γιατί οι κεφαλαιοκράτε είναι τόσο πολύ υπέρ της μετανάστευσης. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να πω... ότι η οδηγία θα ικανοποιήσει νομίζω όλες τις πολιτικές ομάδες. Καταρχήν η εποχιακή. Εδώ θέλω να κάνω δύο προσθήκες που αφορούν τις συνθήκες την πληρωμή, τη στέγαση, την εργασία των εποχιακών. Οι συνθήκες αυτές απασχόλησης θα μπορούσαν να βελτιωθούν εάν η οδηγία προέβλεπε έλεγχο των υπηρεσιών που απασχολούν τους ανθρώπους αυτούς, διότι Αυτές ευθύνονται για τις απαράδεκτες συνθήκες εργοδότησης τους. Μερικοί προσλαμβάνονται από τις χώρες προέλευσης τους, άλλοι στη χώρα όπου έρχονται. Επίσης θα ήθελα να πω κάτι που ίσως αντιτίθεται στην θέση της ίδιας μου της ομάδας αλλά που είναι σημαντικό για τις νέες χώρες μέλη. Με την κρίση και την ανεργία πολλοί εργαζόμενοι θα ήταν πρόθυμοι να εργαστούν εποχιακώς σε χώρες που έχουν ισχυρότερες οικονομίες από τη δική τους. Αυτό μην το ξεχνάμε μπορεί να πληρώνονται λιγότερο αλλά η απασχόληση αυτή είναι κάτι για αυτούς καλύτερο από την ανεργία. Ευχαριστώ. Παπα-Νικολάου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να ξαναευχαριστήσω τον κύριο Μωράης για την εργασία του, για τη δουλειά του. Είναι πράγματι συνοπτική και η δουλειά αυτή και υπήρχε η συνεργασία μας πολύ καλή. Είναι πολύ δύσκολο το θέμα και η οδηγία και όπως είπαν και άλλοι, εδώ δεν πρόκειται για αγώνα δρόμου, χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια και ο Κλάβδιος είναι από τους καλύτερους, από τους πιο ικανούς από όλους μας να τρέξει μαραθώνιο. Κάναμε διαβουλεύσεις καθόλη αυτή την περίοδο. Σήμερα έγινε η τελευταία μας συνεννόηση πριν έρθουμε εδώ και θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους συναδέλφους από την Επιτροπή Απασυχόλησης. Είναι πολύ δύσκολο ξαναλέω. Όλοι είχαμε τα αιτήματά μας και τα ενδιαφέροντά μας. Δεν θέλω να επαναλάβω ποια είναι η θέση της ομάδας μου, αλλά απλώς να τονίσω το θέμα της, του κινδύνου κατάχρησης της οδηγίας αυτής. Είναι κάτι πολύ σημαντικό για μας. Αυτά τα προβλήματα στην Ευρώπη που αφορούν την παράνομη μετανάστευση και την πολιτική που πρέπει να εφαρμόσουμε για να την αντιμετωπίσουμε Έχουμε τις διαπραγματεύσεις για το άσυλο, περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματά τους. Η συζήτηση αυτή των εποχιακών συνδέεται και με όλες τις άλλες διαπραγματεύσεις που ανέφερα και θέλω να θέσω ένα ερώτημα προς την Κομισιόν. Η Κομισιόν και το Συμβούλιο πιστεύουν ότι το άνοιγμα της αρχικής πρότασης και προς ανθρώπους που ήδη διαμένουν νόμιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κάτι που μπορεί να γίνει δεκτό μέσα στα πλαίσια της οδηγίας. Μπορούμε δηλαδή να συνδυάσουμε τους κανόνες που ισχύουν για το άσυλο, για τους αιτητές ασύλου και την περίοδο που θεωρούμε ότι πρέπει να θεσπίζεται μέχρι να ληφθεί η απόφαση. Μπορούμε λοιπόν λέγω να συνδυάσουμε το θέμα, το πρόβλημα αυτό με την πρόταση που κάνανε μερικές πολιτικές ομάδες για αυτή την έκθεση. Συνοψίζοντας θα έλεγα ότι Είμαστε αισιόδοξοι ότι φτάνουμε στο τέρμα της διαδικασίας και θέλω ακόμη μια φορά να ευχαριστήσω τη Γραμματεία και όλους τους συναδέλφους για τη συνεργασία που είχαμε. Φοβόμασταν ότι η έκθεση θα ήταν ακόμη πιο δύσκολη, αλλά χάρη στις προσπάθειες όλων και κυρίως του ζηγητή, διευκολύνθηκαν τα πράγματα. Ευχαριστώ. Λοιπόν, τώρα ακούσαμε τις απόψεις των Ευρωβουλευτών. Άρα ώρα είναι να επανέλθουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μετά στο Συμβούλιο. Καταρχήν ε, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην κυρία Σμιτ. Ευχαριστώ. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Μωράης και τον κύριο Κοφεράτη για την εργασία που έγινε και νομίζω ότι ακολουθεί τη σωστή κατεύθυνση ιδίω βάσει της προτάσεως Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να απαντήσω σε ορισμένα θέματα τα οποία έχουν ε, τεθεί πιο συγκεκριμένα σχετικά με τις άδειε. Είναι ένα τεχνικό θέμα αλλά όταν παρουσιάσαμε την πρόταση εμείς ε, αποβλέπαμε σε αυτούς οι οποίοι ερχόντουσαν για λιγότερο από τρεις μήνες να έχουν μία θεώρηση Σέγγεν και πάνω από τους τρεις μήνες μία άδεια ε, αντί να έχουν άδεια από την πρώτη μέρα το Συμβούλιο όμως τώρα ίσως θέλει να διατηρήσει για τους εποχιακούς εργαζομένους και τις μακροπρόθεσμες θεωρήσεις και να μην υποχρεωθεί να εκδώσει άδειε. Υπάρχουν ορισμένες τεχνικές συζητήσεις που αναφέρονται εις το θέμα της Visa Schengen αλλά νομίζω ότι γενικώ αυτό που είναι πολύ σημαντικό δεν είναι τόσο πολύ το γραφειοκρατικό αν είναι μακροπρόθεσμη θεώρηση ή ε, αδιεργασίας αλλά από την πρώτη μέρα οι εργαζόμενοι να έχουν προστασία και δικαιώματα όπως προβλέπεται στην οδηγία και αυτό είναι βασικό. Επίσης για πρώτη φορά η οδηγία αυτή θα καλύπτει από την πρώτη μέρα τους εργαζομένους διότι εάν υπάρχει μετακίνηση μεταξύ εταιριών αυτό ισχύει μετά από τρεις μήνες αλλά επειδή εκεί ε, έρχονται για μικρότερες περιόδους γι' αυτό θέλαμε να είναι καλυπτημένοι από την πρώτη μέρα και το θέμα των θεωρήσεων περιέπλεκε περαιτέρω το πρόβλημα. Επίσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήθελε να καλύψει τους εποχιακούς που ερχόντουσαν και ήθελαν να φύγουν και η προσέγγιση αυτή λαμβάνει υπόψη ότι πρόκειται για ένα μέτρο προσωρινό και παροδικό και ε, χρειάζονται και πιο ευρία ε, προστασία. Δεν υπάρχει θέμα επανένωσης οικογενειών. Για μας τα άτομα αυτά είναι άτομα που έρχονται από εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μετά από κάποιους μήνες που θα καθοριστούν στο Κοινοβούλιο θα ξαναφύγουν. Νομίζω όμως ότι έτσι έχω απαντήσει στα βασικά θέματα και σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ε, φαίνεται ότι έχει πέσει η αυλαία, ελπίζω να μην είναι η τελική αυλαία. Ε, κυρία Σκύβα, εκ του Συμβουλίου, ευχαριστώ. Εν συντομία, να απαντήσω σε ορισμένε απορίες και σε σχέση με τι απαντήσει που έδωσε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για, τις... για το αν θα δίνονται θεωρήσεις ανάλογα, από... ανάλογα με τη διάρκεια τη διαμονή. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι τα δικαιώματα θα είναι ίδια. Σε καμία περίπτωση δεν θα κάνουμε διαφοροποίηση, γιατί διαφοροποιημένη μεταχείριση ε, αποκλείεται εδώ, γιατί διαφοροποιημένη μεταχείριση και διακριτική μεταχείριση είναι απαράδεκτες. Τώρα, ούτε αυτά που αναφέρθηκε από τον προλήσατε συζητήθηκαν στα πλαίσια των εποχιακά οργαζομένων. Νομίζω ότι είναι ξεχωριστά αυτά τα ζητήματα γιατί οι ευρωβουλευτές επειδή ασχολούνται με και θέματα ασύλου ε, ίσως συγχαίουν μερικά θέματα, αλλά εμείς θα προτιμούσαμε αυτά τα θέματα ασύλου να τα διαχωρίσουμε πλήρως από τα θέματα της εποχιακής απασχόλησης. Ευχαριστώ. Thank you. Σας ευχαριστώ. Κύριε Ισηγητά, κύριε Μωράης, θέλετε να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση με τελικά σχόλια. Έφτασε ήδη καθυστερημένο, να μην παρατείνουμε λοιπόν περαιτέρω τη συζήτηση. Ευχαριστώ και πάλι του και ηγετέ για τη συμμετοχή του ε, σε όλε τι συναντήσει. Πάντω είμαι ανοιχτό και πρόθυμο για την ε, διευθέτηση των τελευταίων ε, ζητημάτων που επισήμαναν οι κύριοι Παπα-Νικολάου και ο κ. Παπα-Νικολάου και η κυρία Σαρτζεντίνη. Είμαι ανοιχτό για συμβαστικέ προτάσει και ελπίζω ότι θα καταφέρουμε να σημειώσουμε πρόοδο πριν την ψηφοφορία στην Επιτροπή μας τον Ιανουάριο. Ευχαριστώ πάντως τους συναδέλφους που αναγνώρισαν τις δυσκολίες αυτής της υπόθεσης και τους ευχαριστώ για τη συνεργασία τους. Ευχαριστώ και τη Γραμματεία. Η Ελένη φαίνεται την παρακολουθεί, αλλά μπορείτε να τη διαβάσετε εσείς τις ευχαριστίες μου. Ευχαριστούμε κύριε Μωράης. Μπορούμε να περάσουμε στο τελευταίο θέμα της απογευματινής μας συνεδρίασης. Ε, φαίνεται ότι... πλησιάζουμε στη συνεδρία των συντονιστών. Κανονικά είχε προγραμματιστεί για τις 5, αλλά όπως ε, θα θυμάστε το πρωί προσθέσαμε τελευταία στιγμή ένα νέο θέμα στην ημερήσια διάταξη, ως τελευταίο θέμα της απογευματινής ημερήσιας διάταξης και καλέσαμε την κυρία Βίξτρομ τη συνάδελφο, να μας ενημερώσει για την ε, αποστολή της αντιπροσωπείας ε, στη Σικελία που έλαβε χώρα από, το, από την 5η 24 έως το Σάββατο 26 Νοεμβρίου. Θα μας κάνει μια έκθεση για τα πεπραγμένα της αποστολής αυτής. Ευχαριστώ. Όταν κατεβάσατε α, την οθόνη, φαντάζομαι οι συνάδελφοι σκέφτηκαν ότι τώρα θα περάσουμε στην φάση της αναψυχής. Όχι, θα σας κάνω μια σύντομη επισκόπηση της ε, επίσκεψης της αντιπροσωπείας μας στη Σικελία και Λαμπεντούσα, πέμπτη με Σάββατο την προηγούμενη εβδομάδα, πριν από λίγες μέρες. Η αντιπροσωπεία μας απαρτιζόταν από 10 μέλη, το Σάιμον Μπουσουτήλ, τη Βερονίκ Ματιέ, το Γιώργο Παπα-Νικολάου ε, και το Σαλβατόρια Κολίνο από το ΕΛ, και την Τάνια Φαγιόν, τη Ρίτα Μπορσελίνο και τη Ροζάρια Κροτσέ, το Ροζάριο Κροτσέτα από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Judith Αργεντίνη από του πράσινου, ο Κυριάκος Τριανταφυλλής από την ΚΟΕ και υποφαινόμενη από την Άλντε, που μου και επικεφαλή τη αντιπροσωπεία. Θα ήθελα καταρχήν να σα πω ότι είχαμε προετοιμάσει αυτή την αποστολή σε συναντήσεις που είχαμε με μη κυβερνητικέ οργανώσει, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Frontex, με την ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ, με την οργάνωση Save the Children και πολλέ άλλε οργανώσει. Θα ήθελα να σας εκθέσω μερικές ε, σύντομε εντυπώσεις για κάποιες επισκέψεις που κάναμε. Όχι από όλες τις επισκέψεις. Καταρχήν επισκεφτήκαμε το Centro de Identificazione και Expulsione, το κέντρο κράτησης ε, στο Τράπανη, κράτηση και απέλασης. Βλέπετε ότι πρόκειται για ένα νέο κτίριο που εγκαινιάστηκε το περασμένο Ιούλιο. Είναι από τα πιο καινούργια κτίρια της Ιταλίας και μάλιστα σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε ως κέντρο ε, κράτησης ε, με χωρητικότητα 250 ατόμων, 178 φιλοξενούνταν όσο ήμασταν εκεί και 140 από αυτούς ε, ήταν ετούντες άσυλο. Ε, δεν ε, κρατούνται εδώ ανηλικοί και 90% των α, φιλοξενωμένων ήταν την ίση. ημέρη είναι προθεσμία για την ακρόαση με την Επιτροπή, αλλά τελικά διαπιστώσαμε ότι περίμεναν ένα μήνα και για να εξεταστεί η υπόθεσή τους. Το κέντρο φαίνεται να πληρεί ε, τις προϋποθέσεις, ε, ε, λειτουργεί αποτελεσματικά, μοιάζει με φυλακή και η παρουσία των ετούντων άσυλων στο κέντρο ε, κράτησης ε, χρήζει περαιτέρω εξέτασης, γιατί φαίνεται ότι η τελική νομοθεσία δεν επιτρέπει ε, απομάκρυση τον τον άσυλο σε μια πιο ανοιχτή δομή, σε ένα πιο ανοιχτό κτίριο που θα αποτελούσε ίσως καλύτερη, ε, ε, καλύτερο τόπο διανυκτέρευσης και παραμονής τον άσυλο παρά ένα κτίριο που θυμίζει φυλακή. Συγγνώμη, ας επιστρέψουμε στην προηγούμενη διαφάνεια. Μην κοιτάτε την επόμενη. Ακούστε λοιπόν. Ε, κατόπιν μεταβήκαμε στην Κάρα, που είναι ένα ανοιχτό κέντρο υποδοχής, στο Τράπανη και πάλι. Γιατί από την Κάρα δεν έχω φωτογραφία, από το κέντρο της Κάρα. Πρόκειται για ένα ανοιχτό κέντρο για ετούντες άσυλο. Οι άνθρωποι εκεί κυκλοφορούν ε, ελεύθερα, μπορούν να εισέρχονται και να εξέρχονται σε συγκεκριμένα ωράρια. 233 ε, είναι η χωρητικότητα του κέντρου αυτού, με ανώτατο όριο χωρητικότητας 260. Ε, υπάρχουν και μερικές οικογένειες εκεί από την Ιγυρία, τον Μπαγκλαντές, το Πακιστάν την Γκάμπια, Ερυθρέα και λίγη και από την Τουρκία. Ε, μη συνοδευόμενοι ανήλικοι δεν στεγάζονται στο κέντρο αυτό, αλλά αποστέλλονται σε ειδικά κέντρα. Όταν επισκεφθήκαμε το κέντρο αυτό, διαπιστώσαμε ότι η εγκατάσταση χρήση κατεπηγόντως ε, ανακαίνησης, γιατί υπάρχουν προβλήματα στις ε, τουαλέτες, δεν υπάρχουν καζανάκια, δεν υπάρχουν πόρτες, ε, κουρτίνες, είδαμε δωμάτια με στρώματα κατάχαμα, 14 και. Οι συνθήκες υγιεινής ε, ήταν ε, ε, ελεηνές όπως μας ενημέρωσαν οι διαμένοντες παρόλο που το κτίριο καθαρίστηκε λίγο πριν τη δική μας επίσκεψη πάντως οι συνθήκες πραγματικά είναι απάνθρωπες και είναι ανάξιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μεταχειρίζεται έτσι ανθρώπινα όντα τον 21ο αιώνα. Αυτή τουλάχιστον είναι η προσωπική μου γνώμη. Μπορούμε τώρα να περάσουμε στην επόμενη φωτογραφία. Αυτό που βλέπετε εδώ είναι πλοιάρια που έχουν ναυαγίσει από την Τινησία κοντά στη Λαμπεντούσα. Όπως ξέρετε η κατάσταση στην Ιταλία αλλά και στην Ευρώπη ολόκληρη δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί αν δεν ε, λάβουμε υπόψη και την κατάσταση της Λαπεντούσα. Η Λαπεντούσα είναι μικρό νησί, τη της Σικελίας, είναι πιο κοντά στην Τινησία από ό,τι στη Σικελία και είναι η πύλη διόδου της, στην Ευρώπη πολλών μεταναστών που περνάνε τη Μεσόγειο με πλοιάρια, ελπίζοντας ότι θα βρουν καλύτερη ζωή. Στην εικόνα αυτή βλέπετε διάφορα πλοιάρια που έχουν εξοκύλει 8 έχουν έχουν, ε, ε, είχαν απομακρυνθεί από το λιμάνι την παραμονή που θα φτάναμε εμείς από την αρχή του, της δεκαετίας του 2000 έχει αυξηθεί η μετανάστευση προς τη Λαμπεντούζα μέχρι σότου υπεγράφει μία συμφωνία για να υπάρχει επαναπατρισμός στην Λιβύη για τους κατοίκους που ερχόντουσαν από εκεί όπως γνωρίζουμε. Υπήρχε δυνατότητα να παραμείνουν 850 άτομα στη Λαμπεντούζα αλλά αυτό έχει ξεπεραστεί και κατά 200 άτομα κατά εποχές οι οποίοι κοιμούνται έξω, οι συνθήκες ήταν τραγικές και μετά την Αραβική Άνοιξη ε, ξαναξεκίνησε ε, το πρόβλημα μέχρι το Μάιο υπήρχε μια μεγάλη συρροή και μια αύξηση ακόμη κατά 48% ως τον Αυγούστο δηλαδή δυόμιση φορές η δυνατότητα υποδοχής του κέντρου αυτού ήταν ο αριθμός των ατόμων που έφταναν <clears throat> και ορισμένοι ε, το σκαγάνε και ε, ερχόντουσαν στα χέρια με ε, τους κατοίκους της περιοχής. Ήταν η εποχή όπου το λιβικό καθεστώς υποχρέωνε τους τινησίους ε, ε, ε, είτε να, είτε να περιληφθούν στο στρατό και να πολεμήσουν τους επαναστάτες ή με την απειλή όπλου να μπαρκάρουν στα πλοία αυτά και να εγκαταλείψουν τη χώρα. Οπότε το κέντρο της Λαμπεντούζας αποτελείται από 7 κτίρια, εκ των οποίων 3 είναι διοικητικά κτίρια και 4 είναι κοιτώνες και βλέπουμε εδώ ένα από τους τέσσερις κοιτώνες και θα σας δείξω κι άλλον έναν αλλά ουσιαστικά ε, πέντε από όλα τα κτίρια είναι ουσιαστικά ασφαλή. Το κτίριο όμως τώρα έκλεισε από όταν οι Ιταλικές αρχές θεώρησαν ότι δεν είναι ασφαλή λες λιμάνι ε, η Λαμπεντούζα για τους μετανάστες όχι για την αλληλεία ή τους αλλά μαζί με την Τρίπολη είναι το μόνο λιμάνι το οποίο θεωρήθηκε ότι δεν είναι ασφαλές σε όλη τη Μεσόγειο. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει ένας ε, κοινός ορισμός σε ευρωπαϊκό επίπεδο διότι οι ψαράδες φοβούνται ότι εάν ε, βοηθήσουν ε, τους ναυαγούς στη θάλασσα θα χρειαστεί να τους μαρκάρουν και να τους συνοδεύσουν μέχρι τη Σικελία και οι διεθνείς οργανώσεις και ακόμη και η τοπική εκκλησία ο επίσκοπος της Λαμπεντούζα τον οποίο συναντήσαμε δεν είναι ε, ε, ικανοποιημένοι με αυτή τη δήλωση του ανασφαλούς λιμανιού για τους μετανάστες. Όπως σας είπα υπάρχει ε, φοβερή ανθρωποπλημμύρα και όλα αυτά ανέρχονται και πριν την περίοδο της 20 Σεπτεμβρίου αλλά η καταστροφή του καταβλισμού οφείλεται ε, στην αντίδραση της παραπομπής προς το Μιλάνο ή προς άλλες περιοχές και είναι ένα θέμα που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε. Ποτέ δεν μπορείτε δηλαδή να μιλήσετε για μετανάστευση και ε, ε, χωρίς να αναφέρετε τη Λαμπεντούζα. Και εδώ βλέπετε κάτι παπούτσια. Κάποιος άφησε ε, ένα σαφές αποτύπωμα αλλά η Λαμπεντούζα τώρα έχει κλείσει. Και το ερώτημα είναι αν χρειάζεται χρειάζεται ένα κέντρο ε, για τις ε, διαμετακομιστικό και θα αφήσω τώρα τη Λαμπεντούζα, θα αναφερθώ στα ευρωπαϊκά ε, κεφάλαια και τη Frontex. Βλέπετε εδώ το χριστιανικό κέντρο Hope and Charity στο Παλέρμο, δηλαδή ελπίδα και η φιλανθρωπία στο Παλέρμο που έχει και μη, ένα νοσοκομείο και νομίζω ότι ουσιαστικά η Σικελία μπορεί να αποτελέσει στο θέμα του εθελοντισμού παράδειγμα για ολόκληρη την Ευρώπη ε, πράγμα το οποίο ε, αντισταθμίζει κάποιος την ε, σκοτεινή εικόνα που σας έδειξα προηγουμένως. Βλέπετε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ταμείου Αλληλεγγύης από το 2009 ως το 2011 διέθεσε 190 εκατομμύρια ευρώ και επιπλέον ε, μέτρα εκτάκτης ανάγκης 18 εκατομμυρίων ευρώ επιπλέον για τη μεταφορά των ε, μεταναστών από τη Λαμπεντούζα προς ε, την ενδοχώρα της Ιταλίας. Επίσης οι μεταφορές ε, το προσωπικό κόστισε 14 εκατομμύρια και με ένα ε, ένα ελικόπτερο που παρα, περιπολεί πάνω από τη Λαμπεντούζα. Ε, τώρα έχουν μείνει λίγοι, η Frontex δεν συντονίζει τις ε, ε, επιχειρήσεις μεταφορών, μόνο ανέλαβε ορισμένες, ορισμένους επαναπατρισμούς προς την Ιγυρία. Όπως είδατε αυτή ήταν μία σύντομη παρουσίαση και σύντομα θα ετοιμάσω τη γραπτή έκθεση και θέλω να πω ότι οι Ιταλικές αρχές, η ε, Frontex και άλλοι οργανισμοί έχουν συμβάλει γραπτός στα διάφορα θέματα τα οποία έθεσα και θα ήθελα ε, ο απολογισμός να είναι όσο το δυνατόν σαφέστερος και η Επιτροπή μας να έχει πλήρη ενημέρωση. Τώρα στρέφομαι προς ε, τους ε, εκπροσώπους που ήρθαν σε αυτή ε, την αποστολή. Θέλω να τους ευχαριστήσω όλους. Θεωρώ ότι ήταν πολύ επικοδομητική η κίνηση αυτή. Ευχαριστώ για όλα όσα κάναμε όλοι μαζί και για την καλή συνεργασία που είχαμε. Αν κάποιος έχει ερωτήσεις ε, είμαι στη διάθεσή σας για να σας απαντήσω μαζί με τους συναδέλφους. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Βίξτρομ, σας ευχαριστούμε για την παρουσίαση που μας κάνατε, αλλά και για το έργο που επιτελέσατε στην αποστολή. Φυσικά ζητάμε πολύ το λόγο από τα μέλη της αντιπροσωπείας. Ποιος θέλει το λόγο πρώτα, κύριος Μπουσουτήλ. Θέλω απλώς να ευχαριστήσω την Κεκυλία για την ενδιαφέρουσα παρουσίασή της και την ακριβή παρουσίαση αυτών που είδαμε στη Σικελία και στη Λαμπεδούσα. Συμμερίζομαι την άποψή της ότι ήταν πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία αλλά και πολύ συγκινητική γιατί είδαμε όχι μόνο τους μετανάστες αλλά και όσους εργάζονται με αυτούς. Και συμφωνώ ότι η επίσκεψη στο χριστιανικό κέντρο που λεγόταν Hope and Charity που το διοικεί ένα πολύ άγιος άνθρωπος που λέγεται κύριος Κόντι είναι κάτι που δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Όσο για τη Λαμπεντούσα, όπως και, η κεκυλία, Βίξτρο με ξεπλάγει και εγώ που έμαθα από τον εκπρόσωπο του Frontex ότι το τελευταίο πλοιάριο που έφτασε στη Λαμπεντούζα από τη Λιβύη έφτασε στις 17 Αυγούστου. Δηλαδή την εβδομάδα που έπεσε η Τρίπολη. στα χέρια όσων διοικούν τη χώρα σήμερα. Αυτό δεν μπορεί να είναι τυχαίο. Νομίζω ότι δείχνει αυτά που υποψιαζόμασταν, δηλαδή ότι το καθεστώς του Καντάφη ε, εξεβίαζε την Ευρώπη με το θέμα της μετανάστευσης. Είναι πολύ καλό ότι φαίνεται ότι σταμάτησε αυτό το φαινόμενο γιατί οι συνδέσεις Λιβύης Ένωσης Διαθαλάσσης παραμένουν παράνομες και φέτος και μόνο εκατοντάδες ανθρώπων πνίγηκαν σε αυτές τις διαδρομές. Η απάντηση λοιπόν για την προστασία των μεταναστών είναι να μην αναγκάζονται να μπαίνουν σε τέτοια επικίνδυνα πλοιάρια. Βλέπω ότι με βιάζεται να τελειώσω. Α, όχι, α, τότε να συνεχίσω λοιπόν. Ας σταματήσω παρόλα αυτά. Πάντως ήταν πολύ ενδιαφέρον νέο ότι ο δρόμος της Λιβύης από τη 17 Αυγούστου δεν λειτουργεί πια. Βέβαια ήρθαν δύο-τρία πλοιάρια και μετά, αλλά για τα περισσότερα από την Τινησία. Και με τις αρχές, τις Τινησιακές αρχές, θα το λύσουμε τώρα μάλιστα που έχει προχωρήσει τόσο πολύ στον εκδημοκρατισμό της η Τινησία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε κύριε Μπουσούτιλ. Όλους μας μας εντυπωσίασε αυτό που μάθαμε για την αποστολή ότι δεν έφτασαν άλλα πλοιάρια στην Λαμπεδούζα από τη Λιβύη από τις 17 α, από την Τρίπολη ειδικά ναι, τη Λιβύη από ολόκληρη τη Λιβύη όχι μόνο από την Τρίπολη από τις 17 Αυγούστου. Μέχρι σήμερα δεν έχει έρθει πλοιάριο από εκεί. Από τη Λιβύη. Από τη Λιβύη. Μέχρι σήμερα, ε, μέχρι σήμερα. Είναι σωστό αυτό μέχρι σήμερα. Ναι, α, είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό. Λοιπόν, για να συνεχίσουμε. Ο κύριος Κοντσέτα. Ε, κοιτάξτε. Και εγώ θέλω να συγχαρώ την επικεφαλής της αντιπροσωπείας. Υπήρξε καταπληκτική συνήψε σχέσεις φιλικές με όλους και με όσους επισκεφθήκαμε και με μας γιατί κανονικά κανείς κουράζεται σε μια τριήμερη επίσκεψη με σάντουιτς και τέτοια, αλλά αυτή τη φορά όχι. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα επίσκεψη. Και οι συναντήσεις πολύ ενδιαφέρουσες εξαιρετική αντιπροσωπεία και για άλλους λόγους διότι δεν πρωταγωνιστούσαν κυρίως οι ευρωβουλευτές αλλά οι άνθρωποι που ήρθαμε να δούμε εκεί. Συναντήσαμε εκπροσώπους και των αρχών αλλά και τους ενδιαφερόμενους, τους ίδιους τους μετανάστες. Δεν μπορούμε να πούμε ότι η Λαμπεδούσα είναι ανασφαλές λιμάνι. Έχει οριστεί έτσι, αλλά εγώ δεν το δέχομαι αυτό. Αυτό το λιμάνι έχει μακρά ιστορία υποδοχής ξένων. Δεν μπορούμε να, πούμε, να το ορίσουμε έτσι αυθαίρετα ανασφαλές λιμάνι. Ξέρουμε ποια είναι βέβαια η κατάσταση της Λαμπεδούσα. Έχουν κάπως βελτιωθεί τα πράγματα σε ορισμένες χώρες, αλλά στην Τινησία ας πούμε συνεχίζουν οι ταραχές και στην Κάφσα και αλλού. Η Λιβύη κατά κανένα τρόπο δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι χώρα που δια, όπου ο λαός τη διαβιεί ειρηνικά τέλος δεν έχουν λήξει ακόμα όλα αυτά αλλά αυτές οι μαζικές ροές που παρατηρούνται φαίνεται να έχουν κάπως καμφθεί Βέβαια ένα μέρος αντιλαμπεδούσα πάντοτε όπως και στο παρελθόν θα διαθέτει νόμιμη ή παράνομη μετανάστευση γιατί είναι μία πόρτα. Είναι τόσο κοντά στην την Ισία και στην Ιταλία που είναι φυσικό να συνεχίζονται οι κάποιες ροές για νόμιμους ή παράνομους μετανάστες που προσπαθούν να μπουν από εκεί στην Ευρώπη. Όσο για τα κέντρα κράτησης, χρειάζονται βέβαια περισσότερα χρήματα για να βελτιωθούν οι συνθήκες εκεί και συμφωνώ και με αυτά που υπόθηκαν για το τράπανι. Υπήρχαν απαράδεκτες συνθήκες 250 έμεναν εκεί και μας είπαν ότι είναι απαράδεκτες οι συνθήκες. Σε άλλες εγκαταστάσεις ακούσαμε παράπονα για το φαγητό, για τις επαφές με την αστυνομία κλπ. Στο τράπανι όμως όλοι συμφώνησαν ότι οι συνθήκες ήταν απαράδεκτες και Μάλλον αυτό θα το κρύψουν στον Υπουργό Εσωτερικών της Ιταλίας. Ένα γενικό μάθημα που μπορούμε να πάρουμε από την επίσκεψη αυτή είναι ότι υπάρχουν ορισμένες ελλείψεις στην ισχύουσα οδηγία. Παραδείγματος χάρη. Το θέμα της πληροφόρησης. Υπάρχουν σύγχρονα κέντρα, αλλά ας πούμε δεν έχουν τηλεόραση. Δεν έχουν τηλεόραση. Και η Επιτροπή μας μπορεί να μπορούσε να κάνει κάτι, να αγοράσει μια τηλεόραση στους μετανάστας. Δεν θα κόστιζε και τόσο πολλά. Θα ήταν πολύ ωραία χειρονομία να προμηθεύσουμε μια τηλεόραση στους διαβιούντες εκεί. Έπειτα το δικαίωμα σε νομική συμβουλή. Δεν θα ήταν καλό να είναι υποχρεωτικό να χορηγείται ένα κατάλογος οργανώσεων που δίνουν νομικές συμβουλές στους μετανάστες και τις μετανάστριες διότι έτσι θα ξέρουν θα ήξεραν που να απευθυνθούν νομικά γιατί στην Ιταλία η νομική συμβουλή είναι δωρεάν άλλο θέμα όσοι ζητούν άσυλο όταν απορρίπτεται η αίτηση και πρόκειται για παιδιά που έχουν έρθει στην ηλικία των 12 ετών καμιά φορά μένουν μέχρι και 6 χρόνια μέχρι να ληφθεί η απόφαση. Τι θα απογίνουν δεν εξαφανίζονται μετά την απόρριψη της αίτηση. Πρέπει λοιπόν να βρούμε βιώσιμες λύσεις για αυτό το θέμα της μετανάστευσης. Όσο για την παράνομη μετανάστευση, φυσικά πρέπει να την αντιμετωπίσουμε. Στη Λαμπεδούζα με εντυπωσίασε ότι αυτοί που μένουν οι κάτοικοι της Λαμπεδούσης ε, τα ίδια ρούχα με τους μετανάστας και ρώτησα τους μετανάστες πού τα βρήκατε τα ρούχα σας και μου είπανε από τα σκουπίδια. σκουπίδια. Ή όχι ακριβώς από τα σκουπίδια αλλά από τα κέντρα μάλλον όπου μαζεύουν πεταμένα ρούχα και είναι απαράδεκτο να δίνονται ορισμένοι, να αναγκάζονται να δίνονται από φιλανθρωπία. Γιατί άνθρωποι είναι και αυτοί, δεν είναι ούτε εχμάλωτοι ούτε κρατούμενοι, είναι αιτητές ασύλου και πρέπει να τους εξασφαλίσουμε τα ορισμένα κριτήρια ζωής, τηλέφωνα, τηλεοράση, έχουν ανθρώπινα δικαιώματα όπως οι μετανάστες και οι μετανάστριες. Α, όταν φτάσουν στην Ευρώπη, όταν φτάνουν στην Ευρώπη πρέπει εκεί να έχουν έναν τρόπο διαβίωσης που να μην, για τον οποίο να μην τρεπόμαστε η κυρία Γκόμς θα φύγει ή θα πάρει το λόγο. Ή... Σύντομα, ε, θα ήθελα να σας πω ότι ε, με συγχωρείτε που δεν μπόρεσα να πάω στην αντιπροσωπεία. Νομίζω ότι έχουν απαντηθεί τα περισσότερα ελετήματα αλλά σχετικά με την πρωτοβουλία των πολιτών που ήταν πολύ ισχυρή επιτόπου. Αντιλαμβάνομαι ότι επιπλέον δεν υπήρχαν πλέον αφήξεις πλοίων μετά τις 17 Αυγούστου. Όλα αυτά λοιπόν μπορούν να θεωρηθούν σαν προηγούμενο και είναι πολύ σημαντικό για όλους μας να δούμε αυτές τις εικόνες και να έχουμε αυτές τις πληροφορίες και σας ευχαριστώ. Ο κύριος Γιακολίνο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε όταν με τον Σιμών Μπουζουτήλ ζητήσαμε σαν μέλη ε, του ΕΛΚ να πάμε στην ε, Λία να δούμε την Λαμπεντούζα και τα άλλα σημεία τα οποία ε, ε, επισκεφθήκαμε ε, ήταν πρωτοφανές. Συμφωνώ με τον Κροτσέτα ότι ήταν μια αληθινή επίσκεψη. Μπορέσαμε να συναντήσουμε διάφορα άτομα τα οποία είχαν φτάσει εκεί προσπαθώντας να επιτύχουν ένα όνειρο ανεκπλήρωτο αλλά ήταν μια αληθινή επίσκεψη ε, και ε, με τη βοήθεια της γραμματείας η αντιπροσωπεία μπόρεσε ε, να διαπιστώσει ότι υπήρξαν ορισμένες δομές οι οποίες δεν ήταν στον ύψος των περιστάσεων και επίσης υπήρχαν ορισμένα θέματα πολύ πιο, πολύ πιο ουσιαστικά τα οποία εξετάζονταν επουσιοδός όπως το καθεστώς των προσφύγων ε, έπρεπε λοιπόν ε, να δούμε πού παραμένουν αυτοί οι πρόσφυγες και όπως είπε και η αντιπροσωπεία της κυρίας Βίκστρομ, ε, ας την ονομάσουμε έτσι, διότι δεν έχει ακόμη καλύψει όλο το στόχο της, εκεί υποτίθεται ότι θα έπρεπε να μείνουν οι πρόσφυγες 48 ώρες και μετά να μεταφερθούν. Δεν μπορούσαν να κάνουν διαφορετικά. Άρα πρέπει να ζητήσουμε από τις Ιταλικές αρχές να, να επαναφέρουν και να τροποποιήσουν το καθεστώς του λιμανιού αφού ανακαινήσουν το κέντρο. Μετά πήγαμε στη Σικελία. Ο Κροτσέτα δεν είναι βέβαια πια ε, ε, νεαρούλης ε, και όλοι καταπονηθήκαμε. Καταφέραμε όμως όμως ε, να πάμε... <clears throat> κυρία Μπορσελίνο, εγώ δεν είπα τίποτα για σας. Είπα για τον κύριο Κροτσέτα μόνο. Είδαμε λοιπόν όλα τα οποία έπρεπε να δούμε και αυτό ήταν ένα πρότυπο προς ε, αντιγραφή διότι είδαμε ε, δύο, δύο κέντρα που είναι διαφορετικά μεταξύ τους και εμείς ε, και αυτό το λέω και στον ε, Σάιμον Μπουζουτήλ, στην κυρία Σαρτζεντίνη και τους άλλους συναδέλφους οι οποίοι ήταν εκεί όλοι αυτοί οι οποίοι συμμετείχουν σε αυτή τη συνεδρίαση ε, έπρεπε να δούμε πώς αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα το οποίο είχαν εκπονήσει μαζί με τα άλλα κράτη-μέλη εφαρμόζεται ότι υπήρχαν ε, χίλιοι ε, πρόσφυγες και 12.000 άτομα τα οποία θα έπρεπε να μπορούν ε, να σωθούν και να αποκατασταθούν στην κοινωνία. Γιατί όχι λοιπόν τώρα έχουμε μία κυβέρνηση τεχνική και ίσως κύριε Πρόεδρε θα έπρεπε ε, να ακούσουμε τις απόψεις της Ιταλικής κυβερνήσεως για να υπάρχει καλύτερη σύνδεση με την Ιταλική κυβέρνηση. Ευχαριστώ. Κύριε Τριανταφυλλίδη, κανονικά τώρα πρέπει να ξεκινάμε τη συνεδρίαση των συντονιστών. Σας θερμό παρακαλώ λοιπόν και εσάς και όλους τους υπόλοιπους ομιλητές που είναι γραμμένοι στον κατάλογο να κάνουν ό,τι μπορούν και να μην ε, μακρηγορήσουν. Ο κύριος Τρενταφυλλίδης. Θα ήταν αχρίαστη επανάληψη αν περιέγραφα και εγώ αυτά τα οποία έχουμε δει. Θέλω να ευχαριστήσω τη Σισίλια γιατί έκαμε μια πάρα πολύ λεπτομερή περιγραφή και τους άλλους συναδέλφους. Θα σταθώ μόνο σε δύο σημεία που μας εισηγήθηκαν η κοινωνία των πολιτών της Λαμπετούσας και που νομίζω ότι είναι σημαντικά. Το ένα είναι η απέτηση τους όπως ο σταθμός της Λαμπετούσας μετατραπεί σε διαμετακομιστικό σταθμό, δηλαδή να μην δέχεται μετανάστες οι οποίοι να μένουν εκεί για μέρες ε, είτε για να εξακριβωθεί η ταυτότητά τους είτε για να απελαθούν, αλλά να γίνει ένα σταθμός όπου θα τους ε, υποδέχονται, θα τους δίδονται τα πρώτα χρειώδη και να μετακομίζονται μετά σε εξειδικευμένα κέντρα υποδοχής όπου θα γίνεται η έρευνα αν είναι αιτητές ασύλου κλπ. Και το δεύτερο σημείο που ήδη έχει αναφερθεί είναι όπως τερματιστεί ο χαρακτηρισμός του λιμανιού της Λαμπετούσας ως ανασφαλές λιμάνι να γίνει ένα λιμάνι υποδοχής γιατί όπως μας έχει εξηγηθεί εκεί πέρα από αρχαιοτάτων χρόνων γεωγραφικά η Λαμπετούσα είναι στο σταυροδρόμι των ροών μεταναστών και φυσιολογικά οι μετανάστες το πρώτο μέρος που θα πλησιάσουν θα είναι η Λαμπετούσα. Επομένως πρέπει αυτό το λιμάνι να ανοίξει και να γίνει ένας ασφαλισμένος σταθμός υποδοχής. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε. Κύριε Αντζελίλη, παρακαλώ, χρόνου φίδου. Θα είμαι λακωνικότατη. Λυπάμαι που δεν έλαβα μέρος στην ε, επίσκεψη αυτής της αντιπροσωπείας, αλλά γνωρίζω αρκετά καλά την κατάσταση στη Λαμπεντούζα, γιατί μαζί με τον Ερθρό Σταυρό και το Save the Children ήμασταν εκεί το Μάρτιο, στην πιο κρίσιμη στιγμή του προβλήματος. Θα ήθελα πάντως να υπενθυμίσω στα μέλη της Επιτροπής μας ότι μαζί με τον κύριο Γιακολίνο είχαμε καταθέσει την πρόταση ενός πιλωτικού προγράμματος εκ μέρους της Επιτροπής που ε, ε, επελέγε μετά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συμπεριλήφθηκε στο προϋπολογισμό που εγκρίθηκε την Πέμπτη με επίκεντρο τους, ε, τα παιδιά, τους, τους ανήλικους μετά από την εμπειρία που συγκεντρώσαμε στη Λαμπεντούσα, αλλά όχι μόνο, μετά από εμπειρίες που είχαμε και από ε, τις εμπειρίες των μη κυβερνητικών οργανώσεων, αλλά και με δική μας παρουσία στην ε, περιοχή, καταθέσαμε ένα πιλωτικό πρόγραμμα για τους ανηλίκους που έγινε ήδη δεκτό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κύριε Μπορσελίνο, παρακαλώ και εσείς ε, να είστε σύντομοι. Θα ήθελα απλώς να επισημάνω δύο στοιχεία. Καταρχήν, το κέντρο της Λαμπεντούσα δεν είναι αλήθεια ότι ε, έχει αχρηστευτεί το κτίριο, όλοι, έχουν αχρηστευτεί όλες οι εγκαταστάσεις. Μπορεί μερικά κτίρια να υπέσαν βλάβες, αλλά δεν ε, έχει, ε, έχει γίνει χρησιμοποιητό όλο το κέντρο. Θα μπορούσε κάλλιστα με μερικές επισκευές να ανακτήσει το ρόλο που είχε αυτό το κέντρο. Γιατί αρχικά η σκέψη μας ήταν η παραμονή στη Λαπεντούζα να μην ξεπερνούσε τις 48 ώρες. Ήταν απλώς διαμετακομιστικό κέντρο, αλλά είχαμε μια πραγματικά τεράστια ροή μεταναστών που συγκεντρώθηκαν ε, στο κέντρο κάποια στιγμή. Και αφήσαμε τον κόσμο να συνοστίζεται και εντός και εκτός του κέντρου. Η Λαπεντούζα έχει πληθυσμό 4 με 5.000 ανθρώπους και χρειάστηκε να υποδεχθεί ε, πολλές χιλιάδες μεταναστών που υπερδιπλασίασαν, πολλαπλασίασαν τον πληθυσμό του νησιού και μάλιστα το φιλοξενεί είναι θυμισμό σε τέτοια περίπτωση και να υποδεχθεί. Υπήρξε λοιπόν μια έλλειψη οργάνωσης Έφταναν τα πλοιάρια στην ε, Λαμπεντούζα και δεν μπορούσαν να ξαναφύγουν εξαιτία τη κακοκαιρία, μα είπαν. Πώ πώς είναι δυνατόν να ισχύει κάτι τέτοιο. Ιούλιο, Αύγουστο, Σικελία έχουμε πολύ έθριο καιρό. Ακόμα και το, καλοκαί... Ακόμα και το χειμώνα οι καιρικέ συνθήκε δεν είναι τόσο αντίξωε. Εν πάση περιπτώσει, δημιουργήθηκε μία κρίσιμη κατάσταση και μία κατάσταση που ξέφυγε του ελέγχου και χρησιμοποιήθηκε ως πρόσχημα για άλλους λόγους. Σίγουρα η κακοκαιρία επιβραδύνει την διαμετακόμιση, την αποχώρηση των πλοίων, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι την καθιστά αδύνατη. Είχαμε πραγματικά με, μεγάλη απώλεια ανθρώπινων ζώων, απαράδεκτο και πολλές φορές το κέντρο υπέστη βανδαλισμούς έγινα στο Μινέο, για παράδειγμα, σε μια καταπληκτική περιοχή, μια πολύ κακή χρήση του κέντρου. Και μάλιστα εκεί είχαν δημιουργηθεί και, και βίλες για τους αξιωματικούς της Αμερικανικής βάσης που βρίσκεται κοντά στο Μινέο. Το πρόβλημα είναι όμως ότι η διαχείριση αυτού του κέντρου, ήταν μη τι άλλο, ε, ύποπτη ένα συνεταιρισμό, αν δεν κάνω λάθο, το διαχειρίζεται και ε, από ό,τι ξέρω αυτός ο συνεταιρισμός έχει και προβλήματα με τον νόμο, άρα δεν είναι και πολύ αξιόπιστος σε ό,τι αφορά τη διαχείριση. Ερωτώ λοιπόν πώς ε, επιτρέψαμε τόσο παρατεταμένη παραμονή αυτών των ανθρώπων, 8 με 10 μήνες, αντί να μένουν κανονικά 2-3 μέρες σε αυτό το κέντρο. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να ευχαριστήσω και προσωπικά τις ε, ναυτιλιακές ε, αρχές και τις ε, θαλάσσιες περιπολίες, για τις θαλάσσιες περιπολίες που έγιναν, καθώς και για τις σωστικές ενέργειες σε πολύ ακραίες μερικές φορές καιρικέ συνθήκες και ευχαριστώ τους αρμόδιους ε, για τη γενοδορία που επέδειξαν στην εκτέλεση των καθηκόντων τους εκ μέρους του Ιταλικού λαού σύσσωμου. Η κυρία Βικστρόμ παρακαλώ πολύ σύντομα. Ναι, όντως θα είμαι λακωνική γιατί θα δοθεί συνέχεια σε αυτή την επίσκεψη από όλου. Υπήρξαν κάποιες ασάφειες και ανακρίβειες που θα πρέπει να τις διαλευκάνουμε και όπως είπα και προηγουμένω, στην αρχική μου σύντομη παρουσίαση αυτό θα γίνει σταδιακά, γιατί θα πρέπει να διαμορφώσουμε μια τεκμηριωμένη γνώμη για το τι συμβαίνει εκεί. Ευχαριστώ και την Τάνια Φαγιών, γιατί αυτή ήταν η φωτογράφος μας, αυτή τράβηξε τις φωτογραφίες που είδατε, να βοηθήσω και την Ελ Χέλν και τη Μαρία από τη Γενική Γραμματεία, γιατί πραγματικά ήταν ηρωίδες, και να ευχαριστήσω και τους πολιτικούς συμβούλους για την πολύ χρήσιμη συμμετοχή τους και φυσικά να ευχαριστήσω θερμά όλους τους συναδέλφους για την πραγματικά ηρωική συμμετοχή τους στην αποστολή αυτή. Γιατί ξεκινήσαμε κρίνοντας πολύ δύσκολο και σφιχτό το χρονοδιάγραμμα, πολύ φορτωμένο και είπαμε ότι θα χρειαστεί να κάνουμε πολλές θυσίες, τα καταφέραμε και πραγματικά ήταν πολύ καρποφόρα η συνεργασία σε αυτή την αποστολή. Σας ευχαριστώ όλους θερμά. Πριν φύγετε και φαντάζομαι εδώ μπορούμε να ολοκληρώσουμε τη, συνεδρίαση, τη δημόσια συνεδρίαση τη Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών και να περάσουμε στη συνεδρίαση των συντονιστών. Θα ήθελα όμω πριν να κλείσουμε να περιληφθεί στα πρακτικά η εξή παρατήρηση. Από τότε που εξελέγει Ευρωβουλευτή τον Ιούνιο του 2009, για πρώτη φορά α, ε, εξελέγει βραβουλευτή και αισθάνθηκε ιδιαίτερη τιμή με την ανάθεση τη Προεδρία στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών και προσέβλεπα σε στενή συνεργασία με όλου και υπολόγιζα στην καλή συνεργασία και των